I don't have this thing. Okay. Uh, colleagues, I would like to start... Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αρχίσουμε. Σας καλωσορίζω όλους τους παρόντες. Meeting is... Uh, ε, και πρέπει να σας πω ότι μεταδίδεται στο διαδικτύο συνεδρίασή μας. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, η έγκριση του σχεδίου, το οποίο έχετε λάβει. Στις 4 Οκτωβρίου το στείλαμε. Αν δεν έχετε διαφωνίες με την ημερήσια διάταξη, θεωρώ ότι εγκρίνεται. Δεύτερο σημείο, ανακοινώσεις της Προέδρου. Και ως συνήθως θα σας ενημερώσω σύντομα για το τι έχει μεσολαβήσει ε, για το Brexit και θέματα που αφορούν την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Θα θυμάστε ότι την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε ψηφίσει και τώρα ήταν μεγαλύτερη υποστήριξη από την περασμένη φορά, δηλαδή οι περισσότεροι συνάδελφοι που συμφωνούν με τη διατήρηση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Brexit. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι καθώς προετοιμάζαμε το ψήφισμα που συνυπέγραψα και εγώ ως Πρόεδρος Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, συμβάλαμε και εμείς από την πλευρά μας. Ε, ήταν συμβιβαστικό έτσι κι το ψήφισμα. Αλλά αντανακλά και τις ε, δικές μας ε, απόψεις. Επίσης την περασμένη εβδομάδα συνεδρίασε η ομάδα παρακολούθησης για τον τέταρτο γύρο διαπραγματεύσεων με τον ε, Μισελ Μπαρνιέ. Ξέρετε ότι ο τέταρτος γύρος δεν συνοδεύτηκε από την απαραίτητη πρόοδο ή την επιθυμητή για να μπορέσει ο κύριος Μπαρνιέ να κάνει προτάσεις στο Συμβούλιο και εμείς να γνωμοδοτήσουμε περί της επαρκούς ε, πρόοδου που έχει επιτευχθεί. Ας ελπίσουμε αυτή την εβδομάδα να καταλήξουμε ε, σε σχετική ανακοίνωση. Δυστυχώς μαθαίνουμε από τον τύπο Ε, πράγματα που ματαιώνουν τις προσδοκίες μας. Επίσης συναντήθηκα με τον νέο Υπουργό Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Συναντικής Δημοκρατίας Χέλεν Μακέντη ε, και συζητήσαμε θέματα ενδιαφέροντος ε, Brexit. Είχα πολλές συνεδριάσεις επίσης με ε, ευρωπαϊκές αερογραμμές ή αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Δεν είναι δική μας βέβαια αρμοδιότητα, όπως γνωρίζουμε όλοι, αλλά τελικά όλα τα θέματα που άπτονται του Brexit θα μας απασχολήσουν και εμάς. Και υπάρχει μια τάση έτσι να συναντούν όλοι την πρόεδρο και τα μέλη της ε, ΑΦΚΟ, τομείς που θα θυγούν ή θα πληγούν από το Brexit. Και όλα τα μηνύματα που ακούμε από τις αεροπορικές εταιρείες είναι αρκετά ζωφερά. Δεν καθόλου ευχάριστα και εκεί μεγάλα προβλήματα. Επίσης είχα ε, επαφές, δέχτηκα μια επίσκεψη από το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικό και το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών και την αντίστοιχη ομάδα Task Force που είναι αρμόδια για τα θέματα του Brexit και επίσης συναντήθηκα με τέσσερις ή πέντε... Ε, υψηλόβαθμους ε, αξιωματούχους, ε, γενικούς γραμματής Υπουργείων και ε, επικεφαλής δημοσίων υπαλλήλων στη Βόρεια Ιρλανδία από την Βόρεια Ολλανδική κυβέρνηση. Αυτά όλα για το Brexit. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας πω ότι στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ψηφίστηκε ο προπολογισμός του 2018 θα θυμάστε ενδεχομένω ότι είχαμε στείλει και εμείς κάποιες δικές μας τροπολογίες και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από τις 10 τροπολογίες που υποβάλαμε δεν εγκρίθηκαν οι 5 και από τις υπόλοιπες 5 οι 2 εγκρίθηκαν στο σύνολό τους είναι για την εκπροσώπηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο διάλογο με του πολίτε και ε, η δεύτερη τροπολογία για τους Ευρωπαϊκού Δημόσιου χώρου, και οι τρει τροπολογίε για τα πιλωτικά προγράμματα καλύφθηκαν από μία συμβιβαστική. Οι υπόλοιπε πέντε, εκ των οποίων τρία πιλωτικά προγράμματα, δεν υπερψηφίστηκαν στην Επιτροπή Προπολογισμών. Υποθέτω ότι θα τις καταθέσουμε ξανά για την Ολομέλεια αυτές τις τροπολογίες. Τι θα γίνει, χάθηκαν. So now, uh, there, there are, the period for normal amendments is still, uh, still open. Okay, so I just like to sensitize. Λοιπόν, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή. Just a second. Because... No, no, no. They, This are no more amendments. Now we go to plenary. Only groups. groups That's what I'm saying. No, individual members cannot okay. So I would like to those of the colleagues. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρεστε για τα προγράμματα αυτά και τις τροπολογίες, παρακαλείστε να ενθαρρύνετε τις πολιτικές σας ομάδες να υποβάλουν εκ νέου αυτές τις τροπολογίες θα ενημερωθείτε για ποιε είναι οι τροπολογίε που απερίφθησαν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το διάβλο των πολιτικών ομάδων για τι επαφέρετε στην Ολομέλεια. Ε, ατομικά, είτε σε επίπεδο επιτροπή, δεν υπάρχει δυνατότητα να υποβληθούν ξανά αυτέ οι τροπολογίε. Και ένα τελευταίο για το οποίο θα ήθελα να σας ενημερώσω. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών επεξεργάζεται αυτό τον καιρό ένα σχέδιο ψηφίσματος ε, προς απάντηση στο σχέδιο, μάλλον στο έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αρμόδιοι εισηγητές μας είναι ο κύριος Όρμπριχτ και η κυρία Τομά. Το ψήφισμα ε, κατατέθηκε εξ ονόματος Επιτροπής Προπολογισμών. Θα θυμάστε ε, ότι εμείς δεν γνωμοδοτούμε σύμφωνα με τον κανονισμό ε, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εσείς μπορείτε όμως να υποβάλλετε τροπολογίες πριν ε, ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Αυτά ήθελα να σας πω. Τελειώνω εδώ με τις ανακοινώσεις μου. Και περνάμε στο σημείο 3, ε, η συζήτηση για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα έχουμε προβλέψει μισή ώρα για τη συζήτηση αυτή. Ε, γιατί αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε. Ξέρετε ότι δύο συνάδελφοι, ο Πέντρο Σίλβα Περέιρα των Σοσιαλιστών και οι υποφαινόμενοι ε, καταρτίζουμε την έκθεση αυτή. 170 τροπολογίες έχουμε λάβει εμπρόθεσμα 3 Οκτωβρίου έλεγε η προθεσμία και αρχίσαμε να τις μελετάμε, να τις επεξεργαζόμαστε. Να αρχίσω εγώ και θα ζητήσω από τον Πέδρο να συνεχίσει. Με κάποιες εξαιρέσεις, οι περισσότερες τροπολογίες αναφέρονται σε τρία βασικά θέματα. Ε, το θέμα της κοινή επικράτειας, ενός συστήματος βασιζόμενο στο ε, μόνιμο μοντέλο και θέματα νομικής ασφάλειας ή ασφάλειας δικαίου σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του Brexit, πότε θα γίνει αυτό και πώς συνδέεται με τις ευρωπαϊκές εκλογές ε, του 19. Ευρωεκλογές. Σε ό,τι αφορά την κοινή επικράτεια, δύο λόγια μόνο, έχουμε λάβει αποκλίνουσες τροπολογίες, οι περισσότερες καθένας προς την κατεύθυνσή του και στην άποψή του. Υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες που θέλουν να, απαλείψουν, να εξαλείψουν οποιαδήποτε αναφορά στη σύσταση γενιαίας επικράτης και επίσης υπάρχουν και τροπολογίες που προτείνουν αριθμούς για έδρες που θα ενταχθούν σε αυτό το ψηφοδέλτιο 30, 43, 50 για ένα ψηφοδέλτιο επικρατείας ας πούμε για όλη την Ευρώπη ε, με βουλευτές από διάφορες χώρες και ορισμένοι το συνδέουν και με τον αριθμό των ευρωβουλευτών ή με το μέγεθος της χώρας. Όπως καταλαβαίνετε, πού να βρει συμβιβασμό εκεί με τόσο αποκλίνουσες ε, προτάσεις. Οπότε μάλλον τροπολογίες θα ψηφίζουμε τελικώς. Υπάρχουν θέματα επίσης που έχουν να κάνουν με τη νομική βάση. Οι περισσότερες τροπολογίες αναφέρουν το γεγονό ότι συνειδητοποιούμε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τη δημιουργία μιας κοινή ε, εκλογικής επικράτειας ή περιφέρειας. και τον εκλογικό νόμο, αλλά επειδή δεν υπάρχει νομική βάση έχουμε πρόβλημα. Και για την ασφάλεια δικαίου να πω και αυτό. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που προτείνουν να διαγραφεί η αναφορά στην ε, ανασφάλεια δικαίου. Γιατί βάσει του άρθρου 50 μπορεί να παραταθούν οι διαπραγματεύσεις και επίσης ε, μπορεί να ανακληθεί και η επίκληση του άρθρου 50. Θα θυμάστε ότι έγινε πολύ έντονη συζήτηση μεταξύ των ε, νομικών εμπειρογνωμόνων και τελικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα από ό,τι κατάλαβα να αποσυρθεί η ενεργοποίηση του άρθρου 50. Και στο πρώτο μας ψήφισμα του Απριλίου αναφερθήκαμε σε αυτό το ενδεχόμενο και θέσαμε και κάποιες προϋποθέσεις. Υπάρχουν τροπολογίες λοιπόν που δεν λαμβάνουν υπόψη αυτή την αβεβαιότητα που προκύπτει από τα δύο ενδεχόμενα. Εμείς θέλαμε να καλύψουμε όλες αυτές τις αβεβαιότητες και τις ανασφάλειες, αλλά μερικές τροπολογίες δεν το αναγνωρίζουν ως πραγματικότητα ότι δεν υπάρχει πάντα ασφάλεια δικαίου ανάλογα με τις εξελίξεις και έχουν μια άποψη την οποία και προωθούν και στις τροπολογίες. Πέντρο, θες να συνεχίσεις εσύ, παρακαλώ. Okay, thank you. Ευχαριστώ. Κάποια σύντομα σχόλια. Το νόημα είναι να βρεθεί λύση με αυτή την προσπάθεια να έχουμε μια σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμορφούνται με τη συνθήκη της Λισαβόνας, που είναι δίκαιη, λογική και πολιτικά βιώσιμη. Οτιδήποτε και αν κάνουμε, το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ακριβώς ε, δίκαιο, λογικό και πολιτικά βιώσιμο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση από, το σχέδιο, από αυτή του σχεδίου έκθεσής μας. Θα ψηφιστούν και εμείς δεν μπορούμε να τις δεχτούμε ως συνεισφορά για την έκθεσή μας. Ούτε μέσω συμβασμών. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε τροπολογίες που ζητούν καμία ανακατανομή των ε, Βρετανικών εδρών, μείωση του μεγέθους ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτω ώστε να καταλήξει σε μια κλίμακα τελείω διαφορετική από αυτή που πρότειναν οι εισηγητέ. Θα τι ψηφίσουμε αυτέ τι τροπολογίε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει βάση για να φτιάξουμε συμβιβασμού πάνω σε αυτή τη βάση. Και έχουμε και τρία βασικά πολιτικά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε και θα τα συζητήσουμε και εδώ και εν συνεχεία στη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Το πρώτο θέμα αφορά τις επιπτώσεις του Brexit. Μπορούμε να παράγουμε νομοθεσία μέχρι το καλοκαίρι του 2018 θεωρώντας αδεδομένο ότι θα γίνει το Brexit πριν από τις εκλογές του 2019. Μπορούμε νομικός πώς να αποκλείσουμε τη δυνατότητα πιο μακροσκελών διαπραγματεύσεων μετά το 2019 και τις εκλογές. Το σχέδιο έκθεσης δέχεται το status quo. Μέχρι να γίνει νομική πραγματικότητα το Brexit. για λόγους ασφάλειας δικαίου για να δείξουμε σύνεση. Υπάρχουν βέβαια τροπολογίες οι οποίες λένε ότι μπορούμε να παράγουμε δίκαιο εικάζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πια μέλος μετά το καλοκαίρι του 2019 και τα πολιτικά και νομικά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε που απορρέουν. Δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με, την, με τον καταμερισμό των εδρών, όπου έχουμε κάποιες τροπολογίες που ζητούν να υπάρχει ένα μόνιμο σύστημα και να βρούμε έναν μαθηματικό τύπο που θα το εξασφαλίζει. Υπάρχουν τουλάχιστον πέντε διαφορετικοί τύποι σε αυτές τις τροπολογίες προτείνονται δηλαδή, αυτές τι τροπολογίες. Και είναι δύσκολο να δούμε αν υπάρχει βάση για πολιτική συμφωνία με βάση αυτές τις ε, τροπολογίες και, αυτές, και αυτούς τους τύπους. Γιατί έχουμε νέου, νέους τύπους που δεν έχουν ξεζητηθεί ποτέ. Ε, το θέμα της ε, μεθόδου DONT, την, τη μέθοδο την σταθερή, διάφορες μέθοδοι προτάθηκαν σε διάφορες τροπολογίες, τη μέθοδο Cambridge, και θα πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα θέματα για να δούμε αν υπάρχει πολιτική συμφωνία επ' αυτή τη βάση. Για τον καταμερισμό των εδρών υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες που ζητούν κάποιες συγκεκριμένες έντρες για κάποιες ε, χώρες, όχι πολλέ. Θα πρέπει να συζητήσουμε και αυτό το σημείο. Τέλος. Υπάρχουν τροπολογίες που αφορούν την ενιαία επικράτεια, όπως είπε και η Ντανούτα. Έχουμε από τη μία τροπολογίες κατά της ενιαίας επικράτειας και έχουμε και κάποιες άλλες υπέρ της κοινή επικράτειας. Αλλά διαφέρουν μεταξύ τους. Ορισμένοι θέλουν η ενιαία επικράτεια να ισχύσει από το 2018 ή 19 τέλος πάντων, ε, και άλλες τροπολογίε προτείνουν διάφορα μοντέλα της ενιαία αυτής επικράτειας. Τα νούμερα είναι διαφορετικά, ορισμένοι προτείνουν 30 έδρε, άλλοι 43, άλλοι 50. Άλλοι ε, νούμερο εισάριθμο με το, του αριθμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μοντέλα είναι πολύ διαφορετικά σε αυτή την, αυτής της ενιαίας επικράτειας της τροπολογίας που έχουμε. Επίσης έχουμε και μία τροπολογία που λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει αντιστάθμιση. Δηλαδή ότι θα πρέπει να κρατήσουμε τα όρια ανακράτος μέλος που έχουμε στη συνθήκη της Λισαβόνας, ακόμη και αν έχουμε μια ενιαία επικράτεια, κάτι που σημαίνει Αν έχουμε έναν βουλευτή από μια χώρα που εκλεγεί μέσω της ενίας επικράτειας, τότε η, λεγόμενη, η εν λόγω χώρα θα πρέπει να εκλέξει λιγότερους ευρωβουλευτές με τα εθνικά ψηφοδέλτια για τις ευρωεκλογές. Αυτά λένε οι τροπολογίες για την κοινή επικράτεια και για να βρούμε συμβιβασμούς θα πρέπει να κοιτάξουμε αυτές τις τροπολογίες για να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε τέτοιες ε, συμβαστικές λύσεις στο σχέδιο έκθεσης. Σας ευχαριστώ ε, εκ των προτέρων. Περιμένω τα σχόλιά σας και τώρα και μετά στη συνάντηση των σκιωδών ε, εισηγητών beyond το όνομά σα να το χέρι σα. Ο κ. E, mm, e, Είναι διαφορετική η γνώμη μου από τη γνώμη του εισηγητή. Παρακαλώ, ε, πλησιάστε λίγο το μικρόφωνο σας. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι λιγάκι διαφορετική από τη γνώμη των εισηγητών. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να διαιρέσουμε τις έδρες που χειρεύουν μετά το, που απελευθερώνται μετά το Brexit. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κρατήσουμε την ε, σημερινή σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι θα είναι μια ενδεδειγμένη λύση που θα επιτρέψει η δουλειά του Κοινοβουλίου μας να γίνει με τρόπο αποτελεσματικό. Αυτές οι έδρες θα μπορούσαμε να τις αφήσουμε για χώρες που θα ενταχθούν αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι ένα αποθεματικό εδρών, που θα το κρατήσουμε κατά μέρο ε, για χώρε που ενδεχομένω θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, ε, επικρίνω λιγάκι ε, αυτή την ιδέα τη ε, υπερεθνική ενία επικράτεια. Συμφωνώ με αυτό που έχει πει ο κύριος Βέμπερ στο ΕΛΚ όταν συζητήθηκε αυτό το θέμα. Ότι, δηλαδή, Όσοι, όσοι συμμετάσχουν σε αυτή την ενιαία επικράτεια θα είναι δηλαδή πιο, θα νομιμοποιούνται περισσότερο να εκπροσωπούν τους Ευρωπαίους. Αυτή η ιδέα ότι έχουν μεγαλύτερη νομιμότητα από του υπόλοιπου που εκλέγονται αλλιώ δεν ισχύει. Η εκλογή των, Ευρωβουλευτών στα κράτη-μέλη δεν, είναι... δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο νόμιμη. Ούτως ή άλλως αυτή η ενιαία ε, επικράτεια θα είναι ένα κατασκεύασμα και είναι πολύ δύσκολο να το, ελέγξει, να το ελέγξουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Νομίζω επίσης ότι δεν θα πρέπει να αναδιανύμουμε αυτές τις ε, έδρες που χειρεύουν μετά τον Brexit. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι κάπως διαφορετικά ερμηνεύω εγώ τις τροπολογίες. 170 τροπολογίες, αν θυμάμαι καλά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση οι τροπολογίες ως προς την ουσία τους. Καταρχάς, για το ζήτημα της νομικής βάσης. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές τροπολογίες. Έχω καταθέσει και εγώ ε, πολλές και κάποιες άλλες ομάδες έχουν καταθέσει ακριβώς ιδέες, τις ίδιες ότι θα γίνει το Brexit, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος και γνωρίζουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συμμετέχει στις επόμενες ευρωεκλογέ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και αυτή είναι και αυτές είναι και οι νομικές συμβουλές που λαμβάνουμε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε το γεγονός αυτό. Και νομίζω ότι αποδυναμώνει και τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το να μην αναγνωρίζετε κάτι τέτοιο στις διαπραγματεύσεις. Εννοώ. Εμείς λοιπόν, ε, όσοι καταθέσαμε αυτές τις τροπολογίες, θεωρούμε ότι πρέπει να αναγνωριστεί αυτό το γεγονός και όλα αυτά τα άρθρα και τις ιτολογικές σκέψεις που εκφράζουν αμφιβολίες ε, για το ε, Brexit. Ε, πρέπει να προετοιμαστούμε για την πραγματικότητα. Το Μάρτιο του 2019 θα υπάρξει αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τον Ιούνιο ευρωεκλογές χωρίς τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει θέμα συμβιβασμού ως προς αυτό. Το δεύτερο που προσπάθησα εγώ να κάνω με τις τροπολογίες είναι να βρεθεί μια λύση με τη φθήνουσα αναλογικότητα. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα είναι βιώσιμο και το οποίο θα ισχύει και για το μέλλον. Δεν μπορούμε να υπάρξει μια σύνθεση του Κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή ξανά που δεν θα βασίζεται σε, σε μια αντικειμενική μέθοδο. Ο σκοπός λοιπόν των δικών μου τροπολογιών είναι να προτείνω ε, τη μέθοδο, το συμβασμό του Cambridge, ε, μια πλήρης φθήνουσα αναλογικότητα, 600, 699 ε, ευρωβουλευτές και ο πρόεδρος, 700 το σύνολο δηλαδή. Μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες αυτού του μαθηματικού τύπου. Νομίζω ότι είναι δίκαιη, φθήνουσα αναλογικότητα. Είναι ένα σύστημα φθήνουσα αναλογικότητα δίκαιο, το οποίο θα μπορέσει να ισχύσει και για τι επόμενε ευρωεκλογέ, ε, μετά από την επόμενη θητεία, όχι μόνο για τη θητεία δηλαδή 19 με 24, αλλά και μετά. Επίσης, για τις, 6, για τις 8 επιπλέον ε, έδρες ε, για να ε, ισχύσουν οι αρχές ε, επί των οποίων ε, οι περισσότεροι συνάδελφοι μπορούσαν να συμφωνήσουν εδώ στην Επιτροπή μας ότι κανένα κρατος μέλος δεν θα έπρεπε να χάσει έδρα στη διάρκεια της διαδικασίας με την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας της θύνουσας αναλογικότητας, δηλαδή αντί να μειώσουμε τον αριθμό των 21 να έχουμε, να χρησιμοποιήσουμε τις 8 για να, για να ισχύσει αυτή η αρχή, μια προσωρινή αρχή κατά τη γνώμη μου και να μείνουν 13, αλλά θα μπορούσε να γίνει αυτό για το 2019 ως 24, ώστε κανένα κράτος μέλος να μην χάσει έδρα. Επίσης, αυτή, αυτή, αυτό το ψηφοδέλτιο το διακρατικό, Γνωρίζετε, η πρόταση του Μακρόν ήταν να υπάρχει φθήνουσα αναλογικότητα και μετά να χρησιμοποιήσουμε όλες τις υπόλοιπες έδρες για ε, διακρατικές ε, λίστες. Αυτή ήταν η πρότασή του. Εγώ ε, υπέβαλα τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και άλλες τροπολογίες ότι αυτά τα ψηφοδέλτια 13, ε, συγγνώμη, 30 εδρών να φτάσουμε δηλαδή στις 730 ε, έδρες στο Κοινοβούλιο κάποια στιγμή, αλλά προσωρινά 738. Νομίζω ότι είναι εύκολο να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό, αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποιες αρχές. Καταρχάς πρέπει να αποφασίσουμε επί ενός μαθηματικού τύπου, για να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα συνεχώς και κάθε πέντε χρόνια. Πρέπει να είναι ε, βασισμένο στη φθήνουσα αναλογικότητα γιατί αυτό είναι ο στόχος μας. Πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό, θα μειώσουμε τον αριθμό ε, όχι κατά πολύ ε, των ε, εδρών του Κοινοβουλίου και το 2019 να υπάρχει μια διακρατική ε, λίστα. Αλλά πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τους σωστούς συμβιβασμούς με τους εισηγητές και με τους κοιόδης εισηγητές στις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε τρει ενότητε, και εγώ να εξηγήσω τι τέσσερις τις πολλές μάλλον τροπολογίες. Αν κοιτάξουμε συνολικά την εικόνα, επιβεβαιώνουν οι τροπολογίε κάτι που φαίνεται και από την έκθεση. Προσπαθεί το κοινοβούλιο να προβληθεί ισχυρό, αλλά δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου κοινέ ε, θέσεις. Αυτό δεν το καταφέραμε και ούτε με το σύστημα των δύο εισηγητών το οποίο προσπάθησα και εγώ να προσβάλλω και να καταρρύψω στα πλαίσια της συζήτηση για τον κανονισμό του Κοινοβουλίου. Οι τροπολογίες τώρα τι δείχνουν όμως. Ότι πολύ περισσότερο ο κόσμος σκέφτεται με κριτήρια εθνικά και λιγότερο κομματικά. Και αυτό είναι κατάφορο όταν συμψηφίζουν ε, ή συνυπολογίζουν τα υπερεθνικά ψηφοδέλτια ή κάποιοι συνάλληλοι με τα εθνικά. Εδώ φαίνεται ε, ότι ο συλλογισμός φτάνει στα όρια του. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο θαραλέοι για την αναθεώρηση του εκλογικού νόμου. Δυστυχώς αυτό δεν το πετύχαμε. Ε, θα πρέπει να βγούμε και να πούμε στον κόσμο ότι Οι έδρες αυτές θα μοιραστούν με τρόπο τέτοιο ώστε να δώσουμε μια ισχυρή πρόταση προς το Συμβούλιο και ό,τι αποφασίσει το Συμβούλιο θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά. Δηλαδή το θέμα που μας απασχολεί ουσιαστικά είναι πώς θα μοιραστούν αυτές οι έδρες. Οι δικές μας τροπολογίες της πολιτικής ομάδας ξεκινούν από την πρόταση των εισηγητών. Ούτε θα φανταστεί κανείς ότι η Γκουε NGL ε, τώρα θα βγει τον τροχό και θα κάνει τελείως διαφορετική πρόταση. Παραμένουμε στο πλαίσιο της έκθεσης. Λοιπόν, η σημερινή κατανομή των εδρών σε πολλές περιπτώσεις παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο και θα πρέπει να το πούμε και θα πρέπει και να το διορθώσουμε. Ε, λοιπόν, πρώτα να αναγνωρίσουμε ότι θέλουμε να το διορθώσουμε και να αυτό δεσμευτούμε. Αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία τώρα του Brexit και ακολουθώ τη λογική των εισηγητών, να περιμένουμε λέτε να ολοκληρωθεί το Brexit, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει μια μέρα όπου η αύξηση ή η μείωση των εδρών θα είναι φυσιολογική, γιατί ε, ε, αλλάζουν και τα δημογραφικά δεδομένα και μετακινούνται και οι πληθυσμοί. Και δεν θα πρέπει να συζητούμε για ένα μόνιμο σύστημα και ερχόμαι στη φθήνουσα αναλογικότητα. Ιδιαίτερα στα μικρότερα κρατημέλη υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν αισθάνεται ο πολίτης ότι εκπροσωπείται και αν εκπροσωπείται. Γιατί κάποια στο Συμβούλιο θέλουν να έχουν πάντα αντισταθμίσματα και αυτό επιδρά και στη δική μας δουλειά. Και είπε ένας Γάλλος συνάδελφος στην ΑΦΚΟ στο Στρασβούργο ότι φθήνουσα αναλογικότητα έχει ε, μια τυπική διάσταση, έχει κάποιες καμπύλες και τα λοιπά και θεωρητικές, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα στα κράτη-μέλη και οι σχέσεις ε, μεταξύ ας πούμε Γαλλίας-Γερμανίας όπως αναφέρεται στο σημείο 11 της έκθεσης. Αυτό θα πρέπει να λυθεί πολιτικά δεν μπορούμε να κρατάμε ισορροπίες ε, και μόνο μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός διόρθωσης των ε, μηχανισμών λήψεων αποφάσεων στο Συμβούλιο. Και τι θα γίνει με το υπερεθνικό ψηφοδέλτιο, πώς θα καταρμηθούν εκεί οι έδρες. Και εγώ, εγώ μιλώ για αναλογική αλλά και ξεκάθαρη ε, αναφορά του, της αρχής don't. Τρίτον, από τις τροπολογίες των συναδέλφων διαβλέπω και εγώ ότι οι περισσότεροι ζητούν πιο ισχυρή πολιτική γραμμή, ιδιαίτερα ε, ως προς το μόνιμο σύστημα που θέλετε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις πραγματικότητες του Brexit και της αναθεώρησης του εκλογικού νόμου, αλλά εάν συμφωνεί η πλειοψηφία στην Επιτροπή μας, θέλω να το εξετάξουμε. Δεν ξέρω αν θα γίνει με συμβιβασμούς ή όχι, δεν είμαι σε θέση να το ε, πω αυτό, γιατί είναι αρκετά δύσκολο, επειδή δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις να βρούμε συμβιβασμούς και νέα γραμμή. Αυτή η προθυμία έχει και όρους και προϋποθέσεις. Υπάρχουν κάποια κατάλοιπα από παλιές εκλογικές περιόδους και εκλογικά συστήματα που επανέρχονται. Η στάθμιση των ψήφων στο Συμβούλιο και εδώ ε, η κατανομή των εδρών βασίζονται στην ίδια ε, βάση υπολογισμού που είναι ο πληθυσμός. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Δεύτερον, μια τέτοια γραμμή δεν θα καθαστεί δυνατή αν προσπαθούμε από τώρα να συνδέσουμε ε, τη θέση του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου με εθνικά κριτήρια και προϋποθέσεις. Και μπορεί να χρησιμοποιούμε ωραίες λέξεις όπως είναι η δικαιοσύνη, η ισότητα κλπ. Και όποιος τα θέλει όλα τελικά δεν πετυχαίνει τίποτα. Να μην είμαστε πλεονέκτες και να μην έχουμε ε, υπερβολικές απαιτήσει γιατί δεν θα βγάλουμε τίποτα. Κατά τα άλλα περιμένω την επικοδομητική συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα ε, στη ρεπουμπλικανική χώρα που είναι η ε, Γαλλία δεν πρέπει να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλικού του βασιλέως, συγγνώμη. Ε, δεν μπορούμε να βάλουμε νομική ασφάλεια εκεί που οι Βρετανοί οι φίλοι μας δεν θέλουν να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Η Τερέζα Μέη, η εκλεγμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, πλέον, είπε ότι το ε, Μάρτιο του 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι μέλος πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είπε κατακάθαρα και εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά ως ευρωβουλευτές ε, να αλλάξουμε τη θέση που επέλεξαν με ελεύθερη βούληση σε ένα δημοψήφισμα πολίτες μια χώρας. Είναι ένα ε, νομικό γεγονός και η Τερέζα Μέη ζήτησε να καταγραφεί αυτό και έτσι ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσει και ο κύριο Φερχόφστα το επενθύμησε αυτό και μα το εξήγησε και ο Μισελ Μπαρνιέ. Μα είπε, μην με υπονομεύετε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων προσπαθώντα να αφήσετε ανοιχτέ πόρτε ε, που δεν είναι ανοιχτέ από κανέναν παρά μόνο από εμά και μόνοι μα βάζουμε τα χεράκια, τα μα και βγάζουμε τα ματάκια μα. Λοιπόν, ε, εγώ θα ήθελα να ζητήσω να μην δημιουργούμε ε, προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Σύμφωνα με τις συνθήκες, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή μας Ένωση το Μάρτιο του 2019. Δεν χρειάζεται να αφήνουμε συνεχώς παραθυράκια, ε, μπορούμε να ε, έχουμε ε, να βάζουμε συνεχώς νέα χρονοδιαγράμματα, όμως υπάρχει το οριστικό χρονοδιάγραμμα του 2019. Ε, δεν θα ήθελα λοιπόν να δημιουργούμε ε, επιπλέον προβλήματα για το θέμα αυτό. Ξεκινώντας λοιπόν από τη σαφή αρχή ότι οι έδρες του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι διαθέσιμες για τις ευρωεκλογές του 2019. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι ρεαλιστής. Είχαμε πει ότι δεν είναι λογικό ε, να πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε από τώρα μέχρι το 2019, αν θέλουμε να μπούμε σε μια διαδικασία αναλογική που θα βασίζεται σε μαθηματικούς υπολογισμούς και μαθηματικούς τύπους, δεν είναι λογικό να θεωρούμε ότι οι χώρες θα δεχθούν να χάσουν έδρες. Δεν είναι δυνατόν να το θεωρούμε αυτό. Οπότε συμφωνώ και με την ε, άποψη που έχει εκφραστεί και στο παρελθόν, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ότι προσπαθούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε βάση μιας αρχής ε, που θα είναι πολύ σαφής να χρησιμοποιήσουμε ένα τμήμα των εδρών για να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε, να υπάρξει μια καλύτερη ισορροπία της αντιπροσωπευτικότητας όλων των κρατών μελών και ε, κυρίως των μικρών και των μεσαίων κρατών μελών. Και γι' αυτό, όπως είπε και ο κύριος Φερχόφστατ, εγώ είμαι υπέρ της χρήσης ε, του power compromise. Νομίζω ότι και εσείς το χρησιμοποιείτε για να υπολογίσετε τις έδρες για το 2019. Μετά όμως, την επόμενη φορά, το 2024, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό τώρα, έχουμε μία ακόμη αρχή ε, που είναι ο συμβιβασμός του Cambridge, η αρχή του Cambridge που δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού με αναλογικό ε, τρόπο ε, και ενδεχομένως για πάντα ή τέλος πάντων όχι για πάντα, για πολλά χρόνια για να το πω έτσι, με αντικειμενικό τρόπο τον αριθμό των εδρών των κρατών είτε προσχωρήσουν άλλα κράτη-μέλη, άλλα κράτη στην Ένωση είτε όχι. Λοιπόν, προτείνω στην πράξη, όπως είπε και ο κύριο Φερχόφστατ, αλλά ενδεχομένω με ένα σύστημα κάπως πιο αντικειμενικό για το 2019, να εφαρμόσουμε το Power Compromise το 2019 και μετά το Cambridge μετά το 2024 για να παραμείνουμε επί αυτής της αρχής ε, να το ε, θεωρήσουμε πια οριστικό, οριστική μέθοδο υπολογισμού από, ε, από εκεί και πέρα. Θα προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω άλλο. Εμείς, ε, εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το υπερεθνικό ψηφοδέλτιο, το έχουμε ξαναπεί άλλωστε, υπήρξε μία πρόταση του Προέδρου Μακρόν, εντάξει δεν είναι βέβαια και Ευαγγέλιο, ε, ότι το 2019 μπορεί να γίνει ένα υπερεθνικό ψηφοδέλτιο και το 2024 να ενισχυθεί αυτό το ψηφοδέλτιο, 50%. Εγώ δεν έχω άποψη ως προς το ποσοστό, αλλά εν πάση περιπτώσει να υπάρχει πάλι μια ρεαλιστική προσέγγιση, να προσπαθήσουμε δηλαδή κάπως να υπάρχει μια εξέλιξη πέρα αυτών των ε, υπερεθνικών ψηφοδελτίων. Δεν ε, πρέπει όμως ε, να συνδέονται τα ψηφοδέλτια αυτά με την εθνικότητα των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτά τα ψηφοδέλτια. Πρόκειται για Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι θα εκπροσωπούν ε, τους πολίτες. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια σχέση μεταξύ των εκλεγμένων, των εθνικών ψηφοδελτίων και την εκπροσώπηση των κρατών μελών που αυτή θα διέπεται από το, την αρχή του Κέμπριτζ όπως είπα προηγουμένως. Καστάλντο ε, δεν είναι εδώ, ο κύριο Άννας δεν είναι εδώ. Πάμε στον κατάλογο των ομιλητών. Σας παραχωρώ δύο λεφτά, όχι παραπάνω. Μετά τα δύο λεφτά θα σας διακόπτω. Κανονίστε ούτω ώστε να πείτε όλα όσα θέλετε να πείτε σε δύο λεπτά. Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα. Έχω 7 ομιλητέ, κλείνω τον κατάλογο. Κύριο Λάινεν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και πολλοί άλλοι πιστεύω και εγώ ότι το Brexit είναι μοναδική ευκαιρία να ανοίξει ένα κεφάλαιο στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν πρόκειται τόσο γρήγορα να έχουμε επόμενη ευκαιρία ελευθερώνονται 73 έδρες που μας διευκολύνουν τη ζωή και για τη φθήνουσα αναλογικότητα, για να τη διαφυλάξουμε έροντας τις ε, αδικίες, αλλά να κάνουμε και κάτι άλλο, το οποίο ζητάει το Κοινοβούλιο μας πάνω από 20 χρόνια. Εκτός από τα εθνικά ψηφοδέλτια στις ευρωεκλογέ, επιτέλους να έχουμε και ευρωπαϊκά ψηφοδέλτια που να επιτρέπονται να συμμετέχουν. Δηλαδή εξευρωπαίζουμε τις ευρωεκλογέ Μπορεί κανείς να θεωρεί ότι αυτό είναι αυτονόητο, αλλά χρειάζεται να το απαιτήσουμε. Δεν έχουμε πραγματικά ευρωεκλογέ, έχουμε 27-28 εθνικέ εκλογέ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν είναι μια μοναδική ευκαιρία να αγωνιστούμε ω Κοινοβούλιο ε, για να συμπεριληφθεί και αυτή η αρχή ε, η δική μα για την κατανομή των εδρών. Ε, στην νομοθετική πρόταση δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Άκουσα ότι μπορούν να υπολογιστούν με βάση το σύστημα DONT, με αντισταθμίσεις. Αυτά όλα δεν είναι του παρόντος ε, οι λεπτομέρειες. Τώρα να συζητήσουμε την αρχή. Και δεν υπάρχει άλλο θεσμικό όργανο που θα αγωνιστεί γι' αυτό, εκτός από το Κοινοβούλιο, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε πολλά κράτη στο Συμβούλιο. Μόνο εμείς μπορούμε να ε, αγωνιστούμε για να αρχίσει η νέα αυτή φάση στο Κοινοβούλιο. Προτείναμε λοιπόν 27 έδρες αναλογία στα 27 κράτη-μέλη το 2019. Τώρα μπορούμε να παίξουμε την κολοκυθιά 30, 40, 50, αλλά το 27 θα αντιστοιχεί σε κάτι. Γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες που αγωνιούν ότι δεν θα έχουμε υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο, θα χάσουμε έδρες, θα τις πάρουν άλλοι. Όλα αυτά είναι για απότερο χρόνο, δεν είναι του παρόντος και περιορίζομαι και σταματώ σε αυτό. Κυρία Ταπερντέρ, δύο λεπτά επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί εισηγητές και αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που φτάσαμε επιτέλους στη συζήτηση των τροπολογιών. Η κατανομή των εδρών ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ των ε, κρατών μελών ε, είναι ένα πολιτικό ευαίσθητο ζήτημα και σημαντικό ζήτημα, ειδικότερα λαμβανομένων υπόψη λαμβανωμένη υπόψη τις σχέσεις που έχουμε με τις χώρες από τις οποίες προερχόμαστε. Το, το μόνο είμαστε το μόνο ε, θεσμικό όργανο που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα, δεν μπορεί να ισχύσει η κατάσταση που ε, ίσχυε το 2013. Χρειάζεται ένα μόνιμο σύστημα κατανομής των εδρών και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για ε, την ε, τρέχουσα θητεία. Επίσης πρέπει να προσπαθήσουμε να αμβλύνουμε τις ανισότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή το σχέδιο έκθεσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Ρουμανία, που έχασαν έδρες το 2013. Δεν νομίζω ότι ήταν σωστό να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει απώλεια εδρών ε, στο μέλλον και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να καταγραφεί. Και αυτή είναι η σωστή χρονική στιγμή να λέμε ότι ε, το 2014-2019 είναι ε, η θητεία αναφοράς, θα ήταν λάθος να το κάνουμε αυτό. Ε, συμφωνώ εν μέρη με την άποψη των εισηγητών, με τη νέα κατανομή, με τη φθήνουσα αναλογικότητα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει απώλεια εδρών για κανένα κράτος μέλος. Παράλληλα όμως, έχω κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με το γεγονός ότι δεν ε, θα είναι σωστή η δημοκρατική εκπροσώπηση αν χώρες ε, με μικρότερο πληθυσμό χάνουν έδρες και οι έδρες αυτές δεν αντικαθίστανται. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ρίτσαρ Κόρμπετ. Δύο λεπτά, Ρίτσαρτ. Δείξε μας ότι οι Βρετανοί καταλαβαίνουν πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος. Ευχαριστώ πολύ και ειδικότερα όπως, εφόσον ε, περνάει ο καιρός, όπως είπε και ο κύριος Μπαρνί. για το ζήτημα αυτό του κατά πόσο η έκθεση πρέπει να προβλέπει ε, τη δυνατότητα ε, ύπαρξης ε, ε, ε, βρετανικών εδρών. Κατά πάσα πιθανότητα το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 20 Μαρτίου του 2019 Στι 29 Μαρτίου του 2019 υπάρχουν όμως τέσσερις ε, ε, συνθήκες υπό τις οποίες δεν θα είναι αυτή η ημερομηνία αποχώρησης. Αν αλλάξει γνώμη το Ηνωμένο Βασίλειο και αποσύρει ε, την ενεργοποίηση του άρθρου 50 ε, και τη σχετική κοινοποίηση, κάτι το οποίο είναι μια πιθανότητα όπως αναφέρει και σχετικό ψήφισμα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης ότι υπάρχει ομόφωνη συμφωνία, το να υπάρχει ομόφωνη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών να παραταθεί η ημερομηνία των διαπραγματεύσεων. Μάλλον απίθανο, κανείς δεν το θέλει αυτό, αλλά μπορεί σε, λίγο, ε, σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να μπορέσουμε να ε, συγκεράσουμε κάπως τις απόψεις μας, να φτάσουμε κοντά σε ένα συμβιβασμό, στο τέλος των διαπραγματεύσεων και συνεπώς μπορεί να υπάρξει τέτοιου είδους πιθανότητα, δεν είναι πολύ πιθανό, αλλά πάντοτε υπάρχει ως πιθανότητα. Τρίτον, να υπάρξει μια συμφωνία σε εύλογο χρονικό διάστημα που θέτει διαφορετική έναρξη ισχύω ε, γιατί η η ημερομηνία αποχώρησης είναι η ημερομηνία της έναξης ισχύω της απόφασης. Εμείς ε, για την ώρα θέλουμε να είναι 29 ε, Μαρτίου του 2019, κάποια στιγμή όμως μπορεί να αποφασιστεί ότι θα είναι μεταγενέστερη αυτή η ημερομηνία. Τέταρτον, να υπάρχει συμφωνία, αλλά να υπάρχει ε, νομική προσφυγή εναντίον της συμφωνίας αυτής, κατά του, ε, ενώπιον του δικαστηρίου. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να γίνει και αυτό. Όλα αυτά τα σενάρια μπορεί να είναι απίθανα σε πολιτικό επίπεδο, αλλά δεν μπορεί να τα αποκλείσει κανένας, οπότε νομίζω ότι η έκθεση θα έπρεπε να το ε, προβλέπει αυτό. Τουλάχιστον τρεις εξημών ε, συμφωνούμε μαζί σου, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε αρκετοί. Μαρτίνα Άντερσον τώρα. Ευχαριστώ τους, τους εισηγητές για την ε, έκθεσή τους. Συμφωνώ με το Χέλμετ και τον Κίθ. Ξέρουμε ποιες είναι οι βρετανικές ε, προθέσεις, παρότι νομικά ε, μπορεί να συμβεί αυτό που λέτε, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αλλά νομίζω ότι τίνω να πιστέψω αυτά που λέει η Βρετανική κυβέρνηση, ότι φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να γίνει ένας διάλογος α, κουφών πάντως. Φυσικά, ε, μία μειοψηφία ε, έχει ξεγελαστεί από τον DUP. Τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, με βάση την τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής έχουν γίνει κάποια πράγματα και αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι στην ε, Βόρεια Ιρλανδία, είναι Ευρωπαίοι πολίτη, πολίτες και λόγω του ε, Ιρλανδικού διαβατηρίου έχουν δικαίωμα να έχουν μάλλον ε, Ιρλανδικό διαβατήριο. Και η τροπολογία 95 ε, λέει πώς θα διατηρήσουμε τη συμφωνία της ε, Μεγάλης Παρασκευής. Δεδομένου το άρθρο 10 της συνθήκης ε, αφορά όλους μας που ζούμε στον Βορρά και αφορά την εκπροσώπησή μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Και εξού και η τροπολογία 144 που θέλει να παρατείνει τον αριθμό των εδρών που δίδονται στην Ιρλανδία, ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι θα έχει επιπτώσεις στην Ιρλανδία τον Brexit, ειδικά σε εμά που λόγω της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, παραμένουμε Ευρωπαίοι πολίτες. Ε, οι τροπολογίες αυτές δηλαδή έχουν σαν σκοπό να διατηρήσουν την ε, συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής σε όλα τα τμήματά της. Άκουσα τι είπε ο Ρίτσαρτ, γιατί όντως κάτι από αυτά που είπε μπορεί να συμβεί. Αλλά μας ε, είπε η Τερέζα Μέη και η κυβέρνησή της με τα ότι φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα πρέπει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια και τη συνεργασία, ε, ειδικά για τη Βόρεια Ιρλανδία. Ε, αυτά και ευχαριστώ. Ο Τζόρτζ Σέπλιν για δύο λεπτά. Συμφωνώ απόλυτα με τον Ρίτσαρντ για το Brexit. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα για την υπερεθνική, το υπερεθνικό, υπερεθνικό ψηφοδέλτιο. Τα έχουμε ξαναπεί εδώ στην Επιτροπή. Το πρόβλημα της ε, λογοδοσίας δεν επιλύεται. Σε ποιον θα λογοδοτούν αυτοί οι ευρωβουλευτές. Ε, πώς θα λειτουργήσει αυτή η λογοδοσία είναι εντελώς ε, ασαφές. Πώς θα υπάρχει επαφή μαζί τους κλπ. κλπ. Πώς θα επιλεγούν αυτοί οι υποψήφοι. Ε, θα γίνει δηλαδή από τους, αυτούς που ασχολούνται με που διαχειρίζονται τα κόμματα, ας πούμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ευρωπαϊκά κόμματα. Και προσοχή, προσοχή, τι επιδιώκεις. Ε, θα ήταν ε, η απότατη ηρωνία ε, να εκλεγούν ε, ευρωσκεπτικιστές στην, ε, στο υπερεθνικό αυτό ψηφοδέλτιο, έτσι. Τώρα, για τον τύπο. Έχω πιστεί ότι κανένας τύπος δεν είναι ιδανικός 100%. Ε, ψάχνουμε τώρα ψιλουστάχυρα. Η εκπροσώπηση είναι ε, καθαρά πολιτικό θέμα, εγγενώς πολιτικό και ο τύπος προσπαθεί να αποπολιτικοποιήσει αυτό το πράγμα, θα δημιουργήσει απογοητεύσεις και θυμό στους πολίτες. Ε, Υπάρχει τεχνοκρατική λύση. Το να χάνει κανεί έδρε είναι επώδυνο, βεβαίω. Εγώ είμαι από την Ουγγαρία, έχουμε χάσει έδρε. Ε, τα κράτη-μέλη θα καταπολεμήσουν μια τέτοια ιδέα, των τύπων δηλαδή, και θα προσπαθήσουν να <clears throat> ε, επαναπολιτικοποιήσουν την, την διαδικασία. Και δίνω και τα υπόλοιπα δευτερόλεπτά μου, τα 20-25 δευτερόλεπτα, στους επόμενους ομιλητές. Ο Ζεγάχ, ευχαριστώ, ε, που μου δίνεις αυτά τα δευτερόλεπτα που σου Τρία σημεία, λέει ο Λαφρίγε, για τον, την εκπροσώπηση και τον αριθμό των ευρωβουλευτών αναχώρα και την προσαρμογή στις δημογραφικές αλλαγές. Έχω κατέξει τροπολογία <clears throat> που σε συνδυασμό ε, με τις άλλες ε, τροπολογίες, τη βλέπω τις άλλες τροπολογίες και ακριβώς θεωρώ ε, ότι καλύπτομαι από τον Γκί Φερχόφστατ. Δεν, δεν μου σημαίνει συχνά. Νομίζω ότι η μέθοδο είναι πολύ πιο απλή, πολύ πιο διαφανή και μπορούμε να μειώσουμε τι αδικίε χωρί να δημιουργούμε καινούριε. Ενώ άλλα συστήματα για να διορθώσουν τι αδικίε νομίζω δημιουργούν μεγαλύτερε αδικίε. Και με αυτή την ε, τροπολογία Γκί θα είμαστε πιο, πιο σαφεί ε, και θα μα δώσει δυνατότητα να πάρουμε και καλέ αποφάσει για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά για τη θέση των Βρετανών που δυστυχώ αποχωρούν. Εγώ δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Έχω, ε, έχω την αίσθηση ότι τα λεπτολογούμε, ψηλολογούμε τόσο πολύ όλα αυτά τα πράγματα. Τι συζητάμε τελικά, το φίλο των αγγέλων. Εγώ το, το συζητούσα με τον Αλάν Λαμασού. Πώς είναι δυνατόν η Βουλή των Κινητήτων ε, να ψηφίσει για να επαναπατρίσει όλο το κοινοτικό δίκαιο, να το έχει στην, ε, να το έχει στη διάθεσή της και αρνείται σε εμά το δικαίωμα να νομοθετούμε για λογαριασμό της τώρα. Πώς λοιπόν επαναπατρίσουν το ευρωπαϊκό δίκαιο και παρόλα αυτά μας δίνουν την αίσθηση ας πούμε ότι ενώ αποχωρήσουν θα εξακολουθούν να παραμένουν πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Ας σταματήσουμε να το ισχυριζόμαστε αυτό. Τρίτο σημείο, για τις, ε, τα υπερεχνικά ψηφοδέλτια. Εγώ είμαι υπέρ της αρχής της δημιουργίας ενός τέτοιου ψηφοδελτίου. Δεν έχω τον τύπο, τον κατάλληλο, την κατάλληλη συνταγή. Ε, ίσως κύριε θα πρέπει να μου δώσετε αυτόν τον ε, μαγικό τύπο που εγώ, εμένα μου διέλαθε, διέλαθε της προσοχής μου. Αλλά ως, ευρωβουλευτές, ως ευρωβουλευτής ε, εκπροσωπώ εγώ το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν εκλεγώ σε μία εκλογική περιφέρεια που βρίσκεται στη Γαλλία, να μην, ε, να μην ξεχνάτε ότι ο κάθε ευρωβουλευτής δεν εκπροσωπεί τους εκλογείς της ε, εκλογικής του περιφέρειας, αλλά το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Είμαι και, ε, εκπροσωπώ και τους Βέλγους, ας πούμε, πολίτες, και τους Γερμανούς και μια άλλη χώρα ως, με τον ίδιο τρόπο που εκπροσωπώ τους εκλογείς της δικής μου εκλογικής περιφέρειας. Αυτό ισχύει για τους ευρωβουλευτές. Δύο χλεφτά κι εσύ. Να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας και να υπενθυμίσω κάτι που είπα και στην αρχή. Ότι είναι σημαντικό να έχουμε τελικά μία δίκαιη και πολιτικά βιώσιμη λύση. Θέλω να πω σε εκείνους που προτείνουν ένα τύπο χωρίς να υπάρξει καμία απώλεια των εδρών μόνο για το 2019, ότι υπάρχει πρόβλημα πολιτικής βιωσιμότητας αυτής της συγκεκριμένης πρότασης, γιατί αυτό σημαίνει ότι για, κάθε, για κάποιες ε, χώρες ότι δεν θα χάσουν έδρες το 19, αλλά θα χάσουν έδρες με συνεχεία. Και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα. Και σοβαρό μάλιστα. Αν το συνδυάσουμε αυτό με την πρόταση για το κοινό ψηφοδέλτιο, όπου κάποιες χώρες, κάποιες μεσαίες χώρες, θα αισθανθούν ότι απειλείται η εκπροσώπησή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αυτά τα δύο σε συνδυασμό θα δημιουργήσουν εκρηκτικό πρόβλημα και δεν θα βρούμε πολιτικά βιώσιμη λύση. Ας κρατήσουμε λοιπόν την αρχή της μη απώλειας εντρών. Νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η αρχή και ας προσπαθήσουμε να δούμε μήπως μπορούμε να πάμε ακόμα παραπέρα σε ό,τι αφορά τις προτάσεις που έχουμε μπροστά μας. Για το κοινό ψηφοδέλτιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σε σχέση με τον εκλογικό νόμο που έχει κολλήσει στο Συμβούλιο εδώ και δύο χρόνια, η Εστονική Προεδρία πήρε πολύ σοβαρά την πρόκληση αυτή και ε, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αφιερώσει σε συζήτηση με τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το θέμα του εκλογικού νόμου. Ελπίζουμε κατά το δεύτερο ήμιση του Οκτωβρίου να λάβουμε πληροφόρηση κατά πόσο έχει υπάρξει καμία εξέλιξη από πλευράς ε, Συμβουλίου. Ε, για μας, ε, αν δεν υπάρχει νομική βάση, μπορούμε μόνο την πρόθεση ε, να εξηγούμε του υπερεθνικού ψηφοδελτίου, κάτι Μόνο αν υπάρχει πλειοψηφία που είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Να σας επιστήσω επίσης την προσοχή στο εξής. Αυτή, αυτός ο μαγικός μαθηματικός τύπος στον οποίο αναφέρεστε αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, πολλές πολιτικές προϋποθέσεις, οι μαθηματικοί τύποι που να ε, πληρούν όλες τις πολιτικές προϋποθέσεις ε, δεν υπάρχουν και πρέπει να το λαμβάνετε και αυτό υπόψη όταν μιλάμε για, την, για το μαθηματικό τύπο όσον αφορά το βιώσιμο σύστημα. Μπορεί να είναι ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται σε βιώσιμες αρχές συμπεφωνημένες που θα βασίζεται σε αρχές διαφορετικές από το μαθηματικό τύπο. Κάτι ακόμη θα ήθελα να σας ε, ζητήσω επειδή το Νοέμβριο στο πρώτο ήμιση του Νοεμβρίου θα γίνουν πολλές συναντήσεις οδών για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε σχέση με την ε, κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσουμε. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από όλες τις πολιτικές ομάδες ε, όταν βρεθεί μια συμφωνία να υπάρξει αν είναι δυνατόν πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο γιατί διαφορετικά δεν ε, θα τα καταφέρουμε πριν από τις εκλογές του 2019. Να κλείσω λοιπόν το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης με τις... Ε, Α, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. θα εξετάσουμε τις τροπολογίες, η τελευταία ελπίζω εξέταση θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα ψηφίσουμε 28 Νοεμβρίου και αυτό κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει ότι θα ψηφιστεί ε, στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο και θα ε, είναι εγκαίρος πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε προβλέψει 40 λεπτά, αλλά θα πρέπει ενδεχομένως ε, να βιαστούμε λιγάκι για το καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο συνεισηγητές ευθύς αμέσως. Ε, Μεσέντες είναι εδώ και οι δύο είναι εδώ. Μεσέντες θα μιλήσει πρώτη. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλοί από εσά άκουσαν ήδη την παρουσίαση τη Κομισιόν στην προηγούμενη συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Ξέρετε, φαντάζομαι, ότι υπάρχει αυτή η πρόταση από την τροποποίηση του ισχύοντος καονισμού και προκύπτει αρχικά αρχικά από ένα ψήφισμα που παρουσίασαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολιτικές ομάδες και που υιοθετήθηκε με πλατιά πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο. Ο στόχος είναι να αυξήσουμε την διαφάνεια, ούτω ώστε οι πολίτες να ξέρουν για ποιον ψηφίζουν, να αυξήσουμε την ε, δημοκρατική νομιμότητα. Το θέμα αυτό συνδέεται πάρα πολύ με το προηγούμενο που συζητήσαμε. Και να ενισχύσουμε την ε, δυνατότητα δράσης εναντίον των καταχρήσεων, καθώς και τη δυνατότητα να ελέγχουμε το πώς δίδονται τα κονδύλια και ενδεχομένως να ανακτούμε τα χρεωστήτως καταβληθέντα. Είναι πολύ σημαντικό το χρονοδιάγραμμα για αυτό το ψήφισμα. Γιατί αν θέλουμε να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί πριν από τις ε, επόμενες ε, ευρωεκλογέ, θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει και ένα τμήμα στο κείμενο που αφορά την καλύτερη λειτουργία της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Θα μιλήσω γι' αυτό. Λοιπόν, στη μεταρρύθμιση που προτείνεται, από τη μία, θέλουμε να σταματήσουν οι καταστάσεις που επέτρεπαν τις ε, καταχρήσεις, να μειώσουμε την πιθανότητα καταχρήσεων. Αυτή τη στιγμή, σε ορισμένε περιπτώσεις, τα μέλη του ίδιου Εθνικού Κόμματος ε, προτείνουν τη δημιουργία ή οδηγούν ε, και είναι η δημιουργή μάλλον ε, διαφορετικών πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, η κατανομή, η διανομή μάλλον των κονδυλίων μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων δεν γίνεται με αναλογικό τρόπο. Όχι επαρκώς αναλογικό τουλάχιστον ε, και δεν λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο της εκπροσώπησης. Ένα μεγάλο κονδύλι, ένα μεγάλο ποσό διαιρείται μεταξύ όλων των κομμάτων ισομερός. Και μόνο το 85% ε, διαιρείται με βάση την πραγματική εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτείνουμε λοιπόν να αυξήσουμε στο στο 95% το κομμάτι που χορηγείται με βάση την πραγματική εκπροσώπηση και μόνο το 5% να μοιράζεται με τον ίδιο τρόπο μεταξύ των κομμάτων ανεξάρτητα από τις ψήφους που παίρνουν δηλαδή. Επίσης η πρόταση προτείνει μια μεγαλύτερη διαφάνεια ανάμεσα Φυσικά η διαφάνεια είναι κάτι το θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτε. Και λοιπόν, ε, η σχέση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα εθνικά κόμματα να είναι μεγαλύτερο η σχέση. Δηλαδή, θα πρέπει ε, τα κόμματα στο site τους να λένε μέσω του λογότυπου τους ε, και του προγράμματούς τους σε ποιο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ε, ανήκουν, ας πούμε. Και στον εκλογικό νόμο που προτείνουμε, ε, προτείναμε ακριβώς ότι πρέπει να ξεκαθαρίζεται από τα εθνικά ευρωπαϊκά κόμματα ε, σε ποιο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ας πούμε, ανήκουν. Ακόμα και όταν δρούν με το συνηθισμένο τρόπο σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να δηλώνουν, ας πούμε, το που ανήκουν. Επίσης, να υπάρχει μεγαλύτερη ε, εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Ε, να το λάβουν υπόψη τους τα κόμματα τα οποία λαμβάνουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία. Παράλληλα, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Να σταματήσουν αυτές οι περιπτώσεις που ανοίγουν πόρτες ούτως ώστε τα κόμματα να καταχρώνται το σύστημα. Επίσης, σημαντικό να τονίσουμε ότι πρόσφατα, μέσω των αλλαγών της νομοθεσίας που εγκρίθηκαν στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου και που τέθηκαν σε ισχύ από το 2017, αλλάζουν κάποια πράγματα, γιατί υπάρχουν μία σειρά από ευρωπαϊκά λεγόμενα πολιτικά κόμματα που δεν κατάφεραν να ε, δώσουν την απαραίτητη τεκμηρίωση, δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα ε, και έτσι δεν δικαιούνται κονδύλια. Τώρα, ο κύριος Βίλαν θα σας πει κάποια πράγματα και αυτός με τη σειρά του και πού μπορεί να υπάρξουν βελτιώσεις αλλά θα ήθελα να σας πω ότι το συζητήσαμε εμεί και προσπαθούμε από τη μία να ξεκαθαρίσουμε τους κανόνες, ούτω ώστε οι στόχοι να μπορούν να υλοποιούνται πολύ πιο εύκολα. Σε ορισμένε περιπτώσει, ε, έχουμε κάποιε αμφιβολίες για τους κανόνες βέβαια. Και δεύτερον, το άλλο που λέγαμε τον κύριο Βίλαντ, είναι το πώς θα επιτρέψουμε στου Ευρωπαίους πολίτε χωρίς να δημιουργήσουμε νέες διαδικασίε να υποδεικνύουν, να δηλώνουν, ας πούμε, καταχρήσεις που είναι εμφανείς στη χώρα τους. Ας πούμε, όταν δεν υπάρχει σεβασμός των βασικών αρχών, ας πούμε, της χάρτας ε, θεμελιωτών δικαιωμάτων. Οι ε, κόμματα τα οποία, ξέρω εγώ, ε, κάνουν ναζιστική προπαγάνδα ή μιλούν, ας πούμε, για την υπεροχή της άριας με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δείχνουν, να υποδεικνύουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρμόδιες αρχές αυτές τις δύο ληστήσεις. Φυσικά θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές μετά να επαληθεύουν αυτά τα λεγόμενα. Οι διαδικασίες θα μπορούν ε, να, χρησιμοποιούν την συνήθη διαδικασία των ε, αιτήσεων, των αναφορών αλλά μπορεί να αλλάξει κατάτικη η διαδικασία από αυτή που ακολουθούμε στις αναφορέ. Γι' αυτό θα χρειαστεί όμως να αλλάξουμε λιγάκι τον εσωτερικό κανονισμό, τους κανόνες κτλ. Είναι τεχνικά θέματα. Το πώς θα επιτρέψουμε δηλαδή στους πολίτες να ε, υποδεικνύουν αυτά τα, αυτές τις δύο ληστήσεις χωρίς να αλλάξουμε εμείς ξανά τους δικούς μας κανόνες. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Όπως σας είπα υπάρχει πρόβλημα χρόνου και θα παρουσιάσουμε ως ονούπο την έκθεση που θα μεταφραστεί εν συνεχεία και η πρόθεσή μας είναι η εξής. Φυσικά η Προεδρία θα μας πει τις ακριβείς ημερομηνίε, αλλά η πρόθεσή μας είναι σε μια έκτακτη συνεδρίαση στην Ολομέλεια, την επόμενη Ολομέλεια του Στρασβούργου, ε, σε μια συνεδρίαση επιτροπής μας λοιπόν έκτακτη, να στο Στρασβούργο τη συζητήσουμε. Συνδέεται επίσης με την προηγούμενη έκθεση και καλό θα ήταν να ψηφίσουμε μέχρι το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια. Εάν θέλουμε, ο μηχανισμός χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, ο νέος αυτός μηχανισμός να τεθεί σε ισχύ. Και κάτι που ξέχασα. Υπάρχει επίσης ένας κανόνας που μειώνει το επίπεδο συγχρηματοδότησης των κομμάτων. και το, το φέρνει στο επίπεδο του 10%. Το υπενθυμίζω αυτό. Εάν θέλουμε να τεθούν σε ισχύ αυτοί οι κανόνες στην επόμενη προεκλογική περίοδο, θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2017 να ψηφίσουμε αυτήν την έκθεση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, Ράινερ Βίλαντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η κυρία Πρέσο παρουσίασε τα περισσότερα και δεν θέλω να τα επαναλάβω εγώ. Θέλω να πω μόνο το εξή. Η νομοθεσία που ισχύει αυτό το καιρό δεν είναι καλή. Εξού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πλήττεται. Αλλά φταίει κιόλα. Έχει πολύ μεγάλο μερίδιο της ενοχής. Υπάρχουν κάποιες τρευλές εξελίξεις λοιπόν που προέκυψαν μετά από πιέσεις και τα λοιπά ε, θέλουμε πριν τις ευρωεκλογέ του 2019 να διορθώσουμε αυτά τα στρεβλά. Τέλη του φθινοπόρου 2018 ε, λίγουν οι προθεσμίες για ορισμένα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήθελε να αλλάξει τίποτα ε, γιατί λέει η ισχύουσα νομοθεσία ότι η αξιολόγηση θα γίνει ένα χρόνο αργότερο. Και ο πρόεδρος Σούλτς και ο πρόεδρος Ταγιάννη πίεσαν όμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει απόφαση και θα πρέπει να τηρήσουμε αυστηρά αυτά που ήδη έχουμε ζητήσει και απαιτήσει μάλιστα. Δηλαδή αυτό είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Δυστυχώς νιώθω ξανά αυτά που συμβαίνουν στο Κοινοβούλιο και στο προηγούμενο θέμα που συζήτησαμε στην ημερήσια διάταξη. Ας πούμε έχουμε τώρα το ρόλο να φτιάξουμε ένα τραπέζι. Και δεν φτιάχνουμε ποτέ ένα τραπέζι. Ε, αλλά κάνουμε διάφορες διαφοροποίησεις και λέμε μπορούμε να φτιάξουμε και ένα τραπέζι με δύο πόδια και μετά όταν πέφτει απορούμε γιατί δεν στέκεται το τραπέζι. Υπάρχουν κάποια πράγματα βασικά που μπορούμε να τα κάνουμε μεθοδικά και γρήγορα και να μην παραφορτώσουμε τη βάρκα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να πούμε στη συζήτηση και ε, πρέπει να σας πω ότι ο ενθουσιασμός στο Συμβούλιο δεν είναι και απεριόριστος. Γιατί αν έχουμε προβλήματα με το Συμβούλιο δεν πρόκειται να προχωρήσουμε στο χρόνο που απαιτείται. Τα περισσότερα τα είπε η κυρία Μπρέσο. Έχουμε ένα ουσιαστικό σημείο, πραγματικά πολύ σημαντικό ε, και χρειάζεται και κείμενο υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι σαφές. Ο αριθμός των βουλευτών που συμμετέχουν σε μια πολιτική ομάδα όταν θέλουμε να υπολογίζουμε ε, τι ποσό τους αναλογεί. Υπάρχουν οι μία εγγεγραμμένοι που δεν ανήκουν σε κόμμα. Αλλά αυτοί θα πρέπει να συνεπολογίζονται στην ε, δύναμη, στο δυναμικό της πολιτικής ομάδας. Προφανώς και όταν υπολογίζεται και το ύψος της χρηματοδότησης, αλλά και όταν υπολογίζεται ε, το γεγονός ε, ότι δημιουργείται, ότι συστήνεται ένα ευρωπαϊκό κόμμα. Εκεί δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται ε, ή αν υπολογίζονται να ανήκουν μόνο σε ένα ευρωπαϊκό κόμμα και όχι σε περισσότερα, γιατί το έχουμε δει και αυτό στο παρελθόν. Λοιπόν, όλα αυτά που έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο να τα ξαναζητήσουμε και με μεγάλη προσοχή, να μην ε, βαρύνουμε πάρα πολύ την πρόταση, να είναι εφαρμόσιμη, να είναι ρεαλιστική, να είναι πρακτική και να έχει και ε, ρεαλιστικές και πραγματικές προοπτικές να περάσει το Συμβούλιο. Έτσι ώστε ε, το Γενάρη, το Φλεβάρι του χρόνου να προλάβουμε και να μην χάσουμε το στόχο μας, να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Όταν έχουμε τέτοιες προτάσεις. καλώ. Ε, καλώς, αλλά προτάσεις για αναβολή θα βρουν αντίθετη και απέναντι την πολιτική μου ομάδα. Θα υπάρξει και επόμενος γύρος ε, στη συνέχεια. Ωραία, σκιώδεις που θέλουν το λόγο. Ο κύριος Μέσσερ Σμιτ από την Ίσια σε Σελίμοβιτς από την ομάδα των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο. Δεν νομίζω ότι η δική μας ομάδα θα είναι εκείνη που θα αντιταχθεί στην πρόταση. Τη θεωρούμε πολύ λογική ε, και σωστή. Κάναμε πάρα πολύ εκτενείς και περιστατωμένες συζητήσεις την περισμένη φορά. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω εγώ. Ε, μερικά πράγματα. Υποστηρίζουμε την ιδέα και την παρατείνουμε και την επεκτείνουμε και στις άλλες διαδικασίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εννοώ αυτή την ιδέα του επικεφαλής του ψηφοδελτίου Spitzenkandidat που ξέρουν οι ε, πολίτες ποιον ψηφίζουν ε, όχι για το κοινοβούλιο μόνο αλλά και για ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινή γνώμη εκλογικού σώματος ή Δήμου με την αρχαία ελληνική έννοια. Τώρα, δεν ξέρω, δεν νομίζω να υπάρχουν προβλήματα. Το ένα είναι η μείωση 15% της υποχρέωσης χρηματοδότησης. Το δεύτερο είναι η αύξηση της ελάχιστης εκπροσώπησης ε, από ένα βουλευτή σε τρεις ευρωβουλευτές για να αποφύγουμε τα μονοκομματικά, μάλλον τα ατομικά κόμματα ενός προσώπου ε, που δημιουργούνται και συστήνονται για να χρηματοδοτούνται και το τρίτο είναι η κατάχρηση ε, πολλαπλών ε, συμμετοχών ευρωβουλευτών σε κόμματα. Κατά τα άλλα συμφωνώ με τους δύο εισηγητές απολύτως και τους ευχαριστώ για την αγαστή συνεργασία και την καλή δουλειά τους. Ευχαριστώ. Σόλτς. Μπορείτε να τα πείτε κι εσείς έτσι τόσο γρήγορα και μεστά. Ε, θα προσπαθήσω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους δύο εισηγητές για τη δουλειά τους. Θα ήθελα να θυμίσω το εξής. Θα πρέπει να γίνεται μια διάκριση εδώ ανάμεσα σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η αναγνώριση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και το δεύτερο είναι η χρηματοδότησή τους. Τεράστια σημασία έχει αυτό, διότι ακόμα και αν δεν έχουν ευρωβουλευτές ούτε έναν, αλλά εκπροσώπους ε, ε, εθνικές ε, συνελεύσεις, βουλές και τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί κάποιος να συστήσει Ευρωπαϊκό Κόμμα. Δεν χρειάζεται να έχει Ευρωβουλευτή. Υπάρχει το δικαίωμα και ελευθερία του συνεταιρίζεστε και τη σύσταση πολιτικών κομμάτων. Το ερώτημα μου τώρα που τίθεται είναι ποια είναι η πολιτική απόδειξη. Εκεί είμαστε πολύ αμυντικοί. όταν δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα μία αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα, όπως είχε ζητηθεί από την προηγούμενη θητεία. Αυτό έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Θα πρέπει να καθίσουμε να δούμε τι θα κάνει η αυτή η αρχή, η ανεξάρτητη ε, και πώς θα αξιολογεί τα κόμματα. Ε, το θέμα της χρηματοδότησης τώρα που είναι διαφορετικό. Καταρχήν, συμφωνώ με τον τρόπο που το προτείνεται, αλλά υπάρχει το εξής πρόβλημα. Αν μειώσουμε τη χρηματοδότηση σε 5% αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι σημαίνει. Ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των βουλευτών δημιουργείται μια ανισορροπία ανάμεσα στα μεγαλύτερα και τα μικρότερα κόμματα. Και αυτό είναι αντίθετο με τις αρχές που έχουμε ε, αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε αυτό, να το ξαναδούμε. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι και τα μικρότερα κόμματα θα έχουν ε, κάποια χρηματοδότηση από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό χωρίς περαιτέρω περικοπές. Γιατί έτσι θα αυξηθούν οι ανισορροπίες και μπορεί να υπάρχει πρόβλημα ε, δημοκρατίας της ίδιας και ως προς την προβολή και τη δραστηριότητα ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Εδώ είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζητήσεις. Και πιστεύω να είμαστε σε θέση να καταλήξουμε στους κανονισμούς αυτούς πριν τις επόμενες ευρωεκλογέ για να μπορέσουν να συμμετέχουν ενεργά τα πολιτικά κόμματα και να υπερασπιστούν και τις κατακτήσεις και τα επιτεύγματα των τελευταίων ε, καιρών και της τελευταίας θητείας, όπως είναι αυτός ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου Spitzenkandidat στα γερμανικά και πρόεδρος αργότερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Χέλμο, το Πασκάλ Ευχαριστώ αντικαθιστώ τον κύριο Καμπράς ε, που έχει δουλειά ε, στην Καταλωνία και δεν θα μπορέσει να έρθει γρήγορα. Πάντως ε, συζήτησα μαζί του χθε και το είπε και ο Χέλμουντ. Θέλω καταρχάς να επανέλθω σε αυτό το σημείο πρώτα. ευχαριστώ τη Mercedes καταρχάς. Συμφωνώ σχεδόν με το 100% των προτάσεών της. Μία δυσκολία έχω με αυτό το σημείο της κατανομής. του κομματιού αυτού που το δίνουμε ας πούμε ισόποσα στα κόμματα. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα που έχουμε στη Γεωργία. Αν αυξήσουμε δηλαδή, αν ξεπεράσουμε τέλος πάντων αυτό το κατόφλι και πάμε από το 85 στο 95, θα έχουμε ουσιαστικά πρημοδότηση ένα εκτάριο. Όσο περισσότερο εκτάρια έχει, τόσο περισσότερα λεφτά θα παίρνει. Για μα αυτό το 15% είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν λέω για μα, ε, εννοώ και για τους ε, πράσινους δεν αλλάζει τίποτα, έτσι, γιατί έχουμε διάφορους ε, εκλεγμένους. Αλλά για την ελεύθερη συμμαχία της Ευρώπης έχουν πολύ λιγότερους εκλεγμένους ε, και αυτό το 15% είναι το 18% του δικού τους ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Το να κόψεις αυτό το ποσοστό και να πας από το 15% στο 5% σημαίνει ότι διάφοροι πούμε, εργαζόμενοι βγαίνουν στην ενεργεία από τη μία στην άλλη. Πρέπει να το εξισορροπήσουμε λιγάκι. Ε, το δίκιο Χέλμουντ. Για μα είναι το μοναδικό πρόβλημα που μα ε, δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί αυτή, αυτό το δεύτερο κόμμα που σα είπα είναι ε, δουλεύουν για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κτλ. Το να χάσει 18% του προπολογισμού του ε, ένα μικρό κόμμα, στην πραγματικότητα το καταδικάζει στην αφάνεια, στην ανυπαρξία. Επομένω, συμφωνώ με το Χέλμουντ, καταλαβαίνω, ξέρω ότι θα τα ακούσει όλα αυτά, θα πρέπει να βρούμε μια λύση για τα μικρά κόμματα. Από το EFTD και το ENF δεν υπάρχουν εκπρόσωποι. Ξαναδείω το λόγο στους εισηγητές. Α, ο Ράινερ. Yeah, yeah, yeah. I just, I just, I just did it. Ναι, μόλις έδωσα λόγο στον κύριο Βίλαντ. Ευχαριστώ. Να πατήσω στο συνάδελφο Σελίμωβιτς, ο οποίος φεύγει. Είπε ο κύριος Σελίμοβιτς ε, κάτι για τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου, Spitzenkandidat στα γερμανικά. Κοιτάξτε, εδώ σας είπα να μην παραφορτώσουμε τη βάρκα. Ε, αυτό, αυτή τη λέξη τη χρησιμοποιούμε και για τον εκλογικό νόμο. Στη Γερμανία υπάρχουν οι επικεφαλείς του ψηφοδελτίου δεν το λέει κανένα νόμος αυτό, ούτε κανένα εκλογικό νόμος. Μπορείς δηλαδή να ορίσει έναν επικεφαλής ή όχι. Σε ορισμένες χώρες έχουμε και μεγάλες επιφυλάξεις κατά του θεσμού αυτού, α πούμε, ή του προσώπου, του επικεφαλής ψηφοδελτίου. Και αν κινδυνεύσει η πρότασή μας, παρόλο που συμφωνούμε, έχω πρόβλημα. Καμία σχέση δεν έχει αυτό με τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Καμία σχέση. Αυτό μπορεί να είναι θέμα του εκλογικού νόμου που κατά δεν είναι. Αυτό αντικατοπρίζει μια πολιτική πραγματικότητα. Ε, ε, με ποιο στυλ πολιτικό προσπαθεί να κερδίσει τους πολίτες ε, για να ψηφίσουν ένα κόμμα. είναι μια ιδέα πούμε, πολιτικού μάρκετινγκ. Δεν έχει καμιά δουλειά στη συζήτηση για τα κόμματα και κύριε Σόλτς, μεγάλα ή μικρά κόμματα. Έγινε η ίδια συζήτηση προηγουμένως για την κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς εξασφαλίζω την ισορροπία ανάμεσα στην αντιπροσωπευτικότητα και την προστασία των μειονοτήτων. Και 5% νομίζω είναι αρκετό για προστασία μειονοτήτων. Και αξιοπρεπέστατο. Γιατί πάντα αυτό το βλέπουμε από τη σκοπιά της μειονότητας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, μου επιτρέπετε, ε, από το χρόνο αγόρευσης στο Κοινοβούλιο. Κάθε πολιτική ομάδα έχει ένα ελάχιστο χρόνο αγόρευσης. Και από εκεί και πέρα, ε, ανάλογα με το μέγεθός της, περισσότερο. Και καμιά φορά προβληματίζομαι κι εγώ και διερωτώ με, πού είναι η δική μου νομιμοποίηση ως βουλευτής μιας χώρας που οι πολίτες έτσι και αλλιώς εκπροσωπούνται με χειρότερο τρόπο αριθμητικά από ότι από μικρότερες χώρες. Πού είναι η δική μου νομιμοποίηση και να βγω να πω στους πολίτες ότι κοίτα να δεις ένα τμήμα του χρόνου αγόρευσης που έχεις ρίξει εσύ στην κάλπη τον εκχωρώ τον χρόνο. Γιατί δεν έχουμε ακόμα αρκετά ε, δικαιώματα για τις μειονότητες. Θα πρέπει να υποχωρούν ακόμα περισσότερο οι μεγάλοι. Και πού είναι το άθροισμα ε, των δικών μας ψηφοφόρων, πού είναι η δική μας ε, νομιμότητα και τα δικαιώματά μας, ε, τα οποία αποκτήσαμε με τις εκλογές, αλλά μετά την εκλογή αποδομούνται συστηματικά. Να μην τα βλέπουμε λοιπόν πάντα από την ίδια σκοπιά. Καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι εδώ οι μικρότεροι θεωρούν ότι η ισορροπία επέρχεται όταν έχουν όλοι τα ίδια, και μεγάλοι και μικροί. Mercedes, thank you, Rainer. Grazie. Mercedes. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τους συναδέλφους, βεβαίως, για τις παρατηρήσεις. Θα συζητήσουμε καλύτερα όταν ε, παρουσιάσουμε το κείμενο, εννοείται. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ότι μειώνοντας το ποσοστό αυτό που πάει ισόποσα σε όλους, που διαιρείται ισόποσα σε όλους, στην πραγματικότητα ε, τη μέρα του λέοντος από αυτό το κομμάτι το παίρνουν οι μεγαλύτεροι. Μεγαλύτερες ομάδες, τα μεγαλύτερα κόμματα. Επίσης, είδαμε ότι υπάρχει μία ε, τάση να πολλαπλασιάζονται τα κόμματα. Εδώ δεν μιλάμε για ομάδες, αλλά για κόμματα, έτσι. Υπάρχει μια ταση να πολλαπλασιαζονται τα Δηλαδή, ένα κόμμα μπορεί να ε, δημιουργήσει δύο, βασικά να, να κλωνοποιηθεί, ας πούμε, για να πάρει περισσότερα λεφτά, έτσι. βλέπουμε ας πούμε ε, καταστάσεις οι οποίες δεν, μπορούν να, δεν πρέπει να γίνονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεδομένου και των νούμερων που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι. Το θέμα είναι να βρούμε μια ισορροπία λοιπόν ανάμεσα στα δύο. Νομίζω λοιπόν ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι αναλογικός προς το βάρος, το ειδικό βάρος που έχει ένα κόμμα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Την παρουσία και την πραγματικότητα που έχει. Γιατί εδώ μιλάμε για πολίτες, για οργανώσεις πολιτών που θα πρέπει να κάνουν μια πολιτική συζήτηση στην Ευρώπη. Διερωτώ με λοιπόν. Ακούμε για κάποια από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα όπου η φωνή τους δεν ακούγεται καθόλου. Ούτε μέσω αδελφών κομμάτων, ας πούμε. Επομένω, το να μην χρηματοδοτούμε τι καταχρήσει μέσω τη δυνατότητα που υπάρχει να πολλαπλασιάζονται αυτά τα μικρά κόμματα, ούτω ώστε να ε, χώσουν το χέρι ας πούμε, σε αυτό το, το κοινό κορβανά, θα πρέπει να το δούμε λοιπόν. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά όταν προκύψει το κείμενο, όταν έχουμε το κείμενο και επί συγκεκριμένων πραγμάτων θα συζητάμε πια. Ο κύριο Σάντεμ ο Διευθυντής της ε, Οργάνωσης των Πολιτικών Κομμάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μερικά πρακτικά ζητήματα θα ήθελα να θέσω σε σχέση με τη διαδικασία. Νομίζω ότι και αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, ώστε το νέο αυτό το σύστημα να δουλέψει σωστά. Νομίζω ότι για τη μετάβαση από το παλιό στο νέο σύστημα χρειάζεται μια σαφής εντολή και μια σαφής διαδικασία για να να γίνει συγκεκριμένη μετάβαση ε, και αυτό είναι κάτι που πρέπει ο νομοθέτης να το αποφασίσει. Υπάρχει μια σαφής νομική βάση και πρέπει επίσης ε, να ε, μην παραμείνουν εγγεγραμμένα όλα αυτά τα κόμματα και ιδρύματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Επίσης μια ένδειξη χρονική πόσο χρόνο θα πάρει αυτή η μετάβαση και επίσης το ζήτημα της αναδρομικής ισχύω ενδεχομένως ε, αυτής της ε, διαγραφής ε, των κομμάτων που επίσης ο νομοθέτης πρέπει να αποφασίσει. Κάτι ακόμη που επίσης αφορά τη διαδικασία Συμφωνούμε με τη νέα πρόταση του άρθρου 27, δυνάμει του οποίου μπορεί τώρα να διαγραφεί ένας ε, ετών όταν έχει υποβάλει λάθος πληροφορίες ε, στην ε, αρμόδια αρχή. Είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει σύμφωνο σε μεγάλο βαθμό. Πιστεύουμε όμως ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί γιατί είναι πολύ ασαφής η διατύπωση και υπάρχουν σαφώς ε, οι παραδείγματα ε, παράγωγης ε, νομοθεσίας της Ένωσης που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να λύσουμε το πρόβλημα. Προτείνω να ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτών. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χρονοδιάγραμμά μας, να σας πω, Επόμενη έκτατη συνεδρίασή μας στις 20... 23 Οκτωβρίου ε, στο Στρασβούργο για να ε, έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε υπόψη και να επεξεργαστούμε περισσότερο τα σχόλια του κυρίου Άνταμ ε, προθεσμοί για τις τροπολογίες 30 ε, Οκτωβρίου, δηλαδή θα έχουμε μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση της έκθεσης και μετά μπορούμε να εξετάσουμε τις τροπολογίες ε, στις 21 Νοεμβρίου στην κανονική μας συνεδρίαση και το Δεκέμβριο τον Ιανουάριο στην, θα γίνει ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Θέλουμε να πάει γρήγορα το θέμα αυτό, γιατί ούτως ή άλλως γνωρίζετε ότι στις 2 Οκτωβρίου αναλάβαμε το θέμα αυτό και το να μην χάσουμε ούτε μία μέρα νομίζω είναι πολύ σημαντικό και επειδή έχει γίνει και μακρά προπαρασκευαστική εργασία πριν από την ε, ε, αρχή της ε, διαδικασίας αυτής. Ελπίζω λοιπόν να πάνε όλα καλά. Ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό της ημερήσιας διαταξής μας και πηγαίνουμε στο 5 που αφορά το ρόλο των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης. Ενδεχομένως να θυμάστε, ο κύριος Ουγιασδόφσκι προετοιμάζει μία έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για το ρόλο των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης και πρότεινε μάλιστα για σήμερα να ακούσουμε εμπειρογνώμονες τους οποίους προσκάλεσε και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα έρθουν εκπρόσωποι από διάφορους φορείς και από πολλά κρατημέλη. Θα ήθελα να αρχίσω δίνοντας το λόγο στον εισηγητή καταρχάς. Ε, κύριε Γιασδόφσκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας. Μισό λεπτό λέει η Πρόεδρος, ε, περιμένουμε λίγο. Ε, αν θέλετε, ελάτε ορισμένοι εδώ στο Προεδρείο να ακούσετε τι θόρυβο κάνετε. Και, καλά, η ακουστική της αίθουσα δεν το συζητώ, αλλά ε, όσοι θέλετε να έχετε ιδιωτικές συνομιλίες, παρακαλώ αποχωρήστε. Τώρα όσοι δεν έχουν ακουστικά δεν με ακούνε και συνεχίζουν να μιλούν και δεν είναι καν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνάδελφοι. Παρακαλώ. Όχι συζητήσει εντός της αιθούς. Ο κύριος ε, έχει το λόγο. Κύριε Ουγεστόφσκι. Έλεγα λοιπόν κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να σας ευχαριστώ πολύ μου ενδιαφέρεστε για το πρόβλημα αυτό ε, το οποίο μας απασχολεί και ευχαριστώ που το γράψατε και στην ημερησία διάταξη. Πρόκειται για το ρόλο των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια κοινή έκθεση της δικής μας Επιτροπής και της Περιφερειακής. είναι και ο κύριος Σόλμπριχτ, ε, εκείνος ο οποίος γνωμοδοτεί στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, παρόν εδώ. Έχουμε και μια ε, μελέτη από το τμήμα μελετών από το Policy Department. Και θέλω να πω πάρα πολύ σύντομα, πριν ακούσουμε τους προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες, δύο λόγια για την έκθεσή μου και το υπόβαθρο, καθώς επίσης και τις πηγές Δύο πράγματα έχουμε εδώ. Τις τελευταίες δεκαετίες πρέπει να πω ότι ο ρόλος των πόλεων έχει ε, αλλάξει στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. η ασφάλεια, οι μεταφορές, ε, μετανάστευση και προς δύο κατευθύνσεις και αστιφιλία και ε, ε, εξωτερική μετανάστευση και ε, ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών. Όλα αυτά είναι θέματα ε, που αφορούν τις πόλεις και ο ρόλος τους αυξάνεται. Ένα δεύτερο στοιχείο ε, είναι να δούμε το δυναμικό που έχουν οι πόλεις, προοπτικά δηλαδή για το μέλλον και ως κοινωνική κινητήρια δύναμη και πώς μπορεί αυτό να προβληθεί στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευρωποίησή τους. Άρα λοιπόν η Ευρώπη είναι μοναδική θα έλεγα διότι δεν υπάρχει πουθενά άλλη ήπειρος στον κόσμο που να έχει τέτοιο δίκτυο αστικών κέντρων ε, τόσο εξέχων και τόσο σημαντικό. Θα πρέπει ταυτόχρονα να υπενθυμίσουμε και ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού και η δική μας συμμετοχή ως Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Αυξάνεται ο ρόλος στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας ενδιαφέρει και μας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο η επιρροή τους και ο ρόλος τους να έχει ένα πραγματικό αντίκτυπο ε, στις δράσεις και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράδειγμα, υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες ε, διαβούλευσης του Συμφώνου του Άμστερνταμ. Αυτή η πλατφόρμα για μένα δεν είναι ούτε ενδεδειγμένη ούτε ικανοποιητική, προσωπική μου άποψη, για να μπορεί να απαντήσει στα υπαρκτά προβλήματα και προκλήσεις. Αυτές οι πλατφόρμες διαβούλευσης τι κάνουν. Ε, είναι ένα δικαίωμα συμμετοχής για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ε, ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει και χρειάζεται μελέτη είναι οι διορθώσεις που γίνονται έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση ε, και μεγαλύτερη των πόλεων στην Επιτροπή των Περιφερειών. Θα δούμε τι θα μας πούν οι εμπειρογνώμονες και οι ειδικοί της Επιτροπής Περιφερειών. Έχουν λοιπόν μεγάλο δυναμικό οι πόλεις και σημαντικό για την αυτονομία τους Και αυτό, όπως είπαμε, είναι καθοριστικό για τη χάραξη της πολιτικής, για την υλοποίηση και για τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί γίνεται ένα διάλογο όπου συμμετέχουν οι πρόεδροι, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, οι διαφόρων αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής. Παράδειγμα, γνωρίζω ότι ο καθηγητής Ματία θα παρουσιάσει ε, μια πρόταση που ξεκινάει από αυτή την παραδοχή. Να δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε τις πόλεις ως ένα κέντρο προβληματισμού και συζητήσεων μεταξύ των πολιτών για να το προβάλλουμε ε, στην ε, λειτουργία και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί λοιπόν ε, γράφονται οι θεσμικοί νεοτερισμοί Πώς μπορούν δηλαδή οι πόλεις να αξιοποιήσουν, να υιοθετήσουν αυτές τις ε, στρατηγικές για να εκτελούν ε, τις ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των υφισταμένων θεσμών ή νέων θεσμών, όπου θεσμικά όργανα θα χρησιμοποιούν αυτό το δυναμικό που έχουν οι πολίτες στην ίδια την πόλη και πώς συμμετέχουν στο γίγνεσθε και στην πολιτική συζήτηση για την Ευρώπη. Αυτά ήθελα να πω τα ολίγα ε, εισαγωγικά. Θα ακούσουμε τις ιδέες ε, που θα μας παρουσιάσουν οι μας και θα τις συμπεριλάβω στην έκθεση. Εκπρόσωπο που έχουμε από την Επιτροπή Περιφερειών, ε, τρεις εμπειρογνώμονες και τον Γιάννα Όλμπρεχ της Επιτροπής Ρέγγι, γιατί γνωμοδοτεί βάσει του άρθρου 54. Ο κύριος Φράνκο Γιάκοπ τώρα παρακαλείται να λάβει το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής των Περιφερειών. Παρακαλώ να σεβαστείτε και το χρόνο σας, 5 με 6 λεπτά. Θα σας ήμουν ευγνώμων. Ευχαριστώ που προσκαλέσατε την Επιτροπή των Περιφερειών στην σημερινή συζήτηση. Το θέμα το αντιμετωπίζουμε με απόλυτη προσοχή και προτεραιότητα. Σε εσά Πρόεδρε, στους συναδέλφους, ε, ε φέρνω τους θερμούς χαιρετισμού του Προέδρου Καρλ Χάινς ε, Λάμπερτς που δεν μπόρεσε να έρθει εδώ σήμερα, γιατί από χθε ξεκίνησε η ολομέλεια τη Επιτροπή των Περιφερειών. Εμεί αντιμετωπίζουμε μια σειρά από προκλήσεων, άνευ προηγουμένου, οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η επίπτωση τη κλιματική αλλαγή, δημογραφικέ αλλαγέ, η ένταξη των μεταναστών, η παγκοσμιοποίηση, η τρομοκρατία, η ριζοσπαστικοποίηση. Η ψηφιοποίηση, η διάδοση των επαναστατικών αυτών τεχνολογιών και αυτές είναι μόνο κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Στην 13 Σεπτεμβρίου ε, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος Γιούνκερ ζήτησε ότι θα ήθελε να δημιουργηθεί μια πιο δυνατή, πιο ενωμένη, πιο δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε αυτό τον στόχο, θέλουμε να υλοποιηθεί και θεωρούμε ότι για να γίνει θα πρέπει να υπάρχει πραγματική εταιρική σχέση με τι ε, πόλει και τι περιφέρειες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να υπάρξει αυτό ο στόχο, θα πρέπει να συνεργαστούμε εμπλέκοντα όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση και τι τοπικέ αρχέ και τις περιφερειακές αρχές προφανώς ε, και όχι με μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω. Εδώ και ε, πολλά χρόνια έχουμε θεωρήσει ότι πρέπει να υπάρχει μια διακυβέρνηση πολυεπίπεδη και είμαστε πεπισμένοι ότι μπορεί να συνεισφέρει στο να λειτουργήσει καλύτερα η Ευρώπη. Ακριβώς γι' αυτό όπως είναι γνωστό, για, ε, ο πρόεδρος και ε, στην ομιλία του ε, μίλησε για τη δημιουργία μιας task force για την επικουρικότητα και την αλογικότητα η δουλειά που κάνει η Ευρωπαϊκή η Επιτροπή των Περιφερειών είναι πολύ σημαντική, ειδικά για ό,τι αφορά ε, την παρακολούθηση τη ε, επικουρικότητα. Και υπάρχει και μια ομάδα παρακολούθηση τη επικουρικότητα και εγώ συνεισφέρω σε αυτήν, ε, συμμετέχω. και νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε με την δουλειά που κάνουμε στην την Task Force. Χθε ο πρόεδρό μα, ο, ο κ. Λάμπερτ, μίλησε, έκανε μια ομιλία για την κατάσταση τη Ένωση και είπε την προοπτική των πόλεων και των περιφερειών και μετά ακολουθήθηκε μια ε, συζήτηση, ακολούθησε συγγνώμη και μια συζήτηση με τον ε, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Τούσκ. Ε, στα πλαίσια μια ευρύτερη συζήτηση και ευρύτερου προβληματισμού, όπου συμμετέχει και η Επιτροπή των Περιφερειών για την κατάσταση αυτή. ο πρόεδρό μα μίλησε για τι βασικέ προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ. Ε, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάνω από 150 εκδηλώσεις, οποίες συμμετέχουμε εμείς, ε, όπως στην εκδήλωση ας πούμε που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τον κύριο Τούσκ για την, ε, τις πόλεις ε, και τις περιφέρειες της Ευρώπης. Ε, όλο και πιο πολύ είναι σημαντικές οι περιφερειακές και τοπικές πολιτικές. Είναι πολύ σημαντικέ για να ενεργοποιηθεί και να εφαρμοστεί και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ειδικά οι περιφέρειες οι οποίε έχουν και νομοθετικέ αρμοδιότητε μέσω ε, περιφερειακών κοινοβουλίων ε, και που εκπροσωπούνται ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο εν συνεχεία αυτές, αυτά τα περιφερειακά κοινοβούλια. Ε, Επίση και το ευρωπαϊκό επίπεδο επηρεάζει τι πόλει και τι περιφέρειες, αλλά και αντίστροφα οι πόλει και οι περιφέρειες θα πρέπει να μπορούν να επηρεάζουν τι ευρωπαϊκέ αποφάσει. Ε, στη συζήτηση στην Ολομέλεια, που μετά την παρουσίαση του Πρόεδρου Λάμπερτ, ο Πρόεδρο Τούσκ δήλωσε ότι η εμπιστοσύνη και η ευημερία της Ευρώπης εξαρτάται από την ζωντάνια των πολεών μας, των περιφερειών μας και των δήμων και κοινοτήτων. Ε, και αυτό απεικονίζεται στην, ε, στο θεματολόγιο, στην ατζέντα της Επιτροπής των Περιφερειών. Εμείς βλέπουμε ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα από κάτω προς τα πάνω, το βλέπουμε σαν προς τα πάνω. Ε, οι πολίτες και εμείς έχουμε ένα σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να παίξουμε στην ευρύτερη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ε, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές γνωρίζουν ποια είναι η, πραγματική, η πραγματικότητα σε τοπικό επίπεδο. Ε, και αυτό μας δίνει μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στους πολίτες και είναι και μια μεγάλη ευκαιρία ταυτόχρονα για την το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ο πρόεδρος Τούσκ μίλησε ε, στα όσα συμφώνησαν ε, στην Πρατισλάβα το Σεπτέμβριο του 2016 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Μια σειρά από συγκεκριμένε δεσμεύσει, ε, ρεαλιστικέ δεσμεύσει, που τις, πολύ επίκαιρε, ούτω ώστε να απαντήσουμε στι ανησυχίε των πολιτών, το κλίμα, η οικονομία, η ασφάλεια κτλ. Είναι απαραίτητο να δράσουμε, ούτω ώστε να μειώσουμε την απόσταση ανάμεσα στη θεωρία και στην πρακτική, ανάμεσα στα λόγια και στα έργα. Ε, ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη το ζουν σε πρώτη γραμμή, σε πρώτη γραμμή πρώτες και καλύτερες οι πόλεις και οι περιφέρειες. Και προφανώς θα πρέπει να συμμετέχουν στην προετοιμασία και στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η ασφάλεια είναι μία από τις βασικές ανησυχίες και τα μελήματα των ευρωπαίων πολιτών σε ένα κόσμο όλο και πιο ασταθή και σε εμά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η τρομοκρατία είναι μια μόνιμη απειλή. Η ριζοσπαστικοποίηση, η απότατη βία, η ακραία βία είναι ε, πράγματα που υποσκάπτουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ε, και εκεί βρισκόμαστε στα χαρακόμματα εμεί οι πόλει και οι περιφέρειες. Χωρί τη συμμετοχή μα δεν μπορούν να υπάρξουν αποτελέσματα. Σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση και εκεί θα πρέπει να ε, υλοποιήσουμε την ένταξη των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό επίση ε, ο ρόλο των πόλεων για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να εφαρμόσουμε την ε, συνθήκη των Παρισίων. Τα τρία τέταρτα των πόλεων, τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων ζουν σε πόλει και σε αστικέ περιοχέ και όλο και περισσότεροι θα ζουν στο μέλλον. Είναι σημαντικό αυτό για την ενεργειακή αποδοτικότητα, τη μείωση του, του διοξιδίου του άνθρακα για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν μεγάλες αστικές αλλαγές, ε, πρωτοβουλίες που γίνονται για το κλίμα και την ενεργεία, το σύμφωνο των δημάρχων. Είναι η μεγαλύτερη τέτοια κίνηση που γίνεται ποτέ, όπου χιλιάδε χιλιάδες τοπικές και περιφερειακές αρχές σε εθελοντική βάση συμμετέχουν σε αυτό το σύμφωνο ε, για να προωθήσουν τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επικράτειά τους. Η ένταξη των μεταναστών, η κοινωνική συμμετοχή είναι διαδικασίε μακροπρόθεσμα που απαιτούν την εμπλοκή όλων των φορέων που έχουν ε, ευθύνη. Τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ε, οι ε, πολίτες φυσικά, οι επιχειρήσεις, οι πάντες. Ο ρόλος ε, της, των πόλεων για την ένταξη μεταναστών φυσικά είναι κρίσιμος. Θα μπορούσα να σας δώσω πολύ άριθμα άλλα παραδείγματα για τη συμμετοχή των πόλεων σε στατικούς τομείς. Ε, εμείς δεχόμαστε υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση με διαφορετικούς τρόπους. Ε, χρηματοδότηση για την προσαρμογή μας στις προκλήσεις κτλ. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίζεται ρητά ο ρόλος των πόλεων μέσω συγκεκριμένων ευρωπαϊκών πολιτικών, ούτω ώστε οι αρμοδιότητέ μα να χρησιμοποιούνται και οι γνώσει μα να ε, χρησιμοποιούνται από το θεσμικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρόλο μα στην ε, πόνηση και εφαρμογή των πολιτικών θα πρέπει να ενισχυθεί. Ελπίζω ότι η Επιτροπή των Περιφερειών θα μπορέσει περαιτέρω να συνεισφέρει στι εργασίε σα για το ρόλο των ε, και ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο να είναι ακόμη πιο έντονος. Και βεβαίως ε, θα διαβάσουμε το σχέδιο αυτού του κειμένου σας και θα, το, θα συνεισφέρουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το πώς μας περιγράψατε όλες αυτές τις προκλήσεις. Ε, ευχαριστούμε επίσης και για τη δέσμευσή σας για συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Ραφαέλ Ματία είναι ο πρώτος προσκεκλημένος μας από ε, το ΖΕΣΟΥΦ ε, από το Τμήμα Πληροφορικής και Διαχείρισης Πληροφορίας. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα ο σκοπός μου είναι να σας εξηγήσω την πρόταση αυτή. Πρέπει να αρχίσω λέγοντας τι δεν είναι αυτή η πρόταση. δεν προτείνει κανένας να κυβερνήσουν τον κόσμο οι δήμαρχοι, ούτε ζητά μεγαλύτερη επιρροή των πόλεων στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μόνο που προτείνει είναι να αποτελούν εταίρους ε, οι πόλεις, να μην είναι μια αποκλειστική λέσχη με μεγαλύτερη επιρροή δεν είναι μια διοικητική οντότητα η πόλη είναι μια λειτουργική οντότητα που έχει το δικό της περιβάλλον, παρέχει υπηρεσίες, είναι πολιτικό κέντρο και κέντρο διαμόρφωσης πολιτικών απόψεων. Ο κεντρικός πυλώνας της πρότασης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αξιοποιήσει το δίκτυο πόλεων της Ευρώπης γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής δεν έχουν τίποτε τέτοιο, ούτε άλλες μεγάλες χώρες του ΟΣΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μοναδική υπ' αυτήν την έννοια. Έχουμε ε, πόλεις ε, που είναι δικτυωμένες, ε, πολλές έχουν ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια, μέσα ενημέρωσης και υπάρχει ανάγκη δημόσια συζήτηση. και πρέπει οι διδάσκοντες να ενθαρρύνουν το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη διαμόρφωση των πολιτικών πεπιθήσεων. Δεν πρέπει απλώς να ε, επαφίεται αυτό ε, στους ε, τοπικούς πολιτικούς. Πρέπει να υπάρχει δημόσια διαβούλευση, δημόσιος διάλογος, έγγραφες διαδικασίες, προφορικός διάλογος επίσης. Στο κάτω-κάτω της γραφής υπάρχουν μικρά πανεπιστήμια σε μικρές πόλεις που μπορεί να έχουν και αυτά μια άποψη για τις πολιτικές της Ένωσης. Αυτή τη στιγμή ε, είναι κάπως παραγνωρισμένες, όμως ε, έχουν το δικαίωμα να πούν κάτι. Μία ε, πόλη ε, όπως η Τεργέστη για παράδειγμα, άλλες μικρές πόλεις πρέπει να μπορούν να εισακούονται και εκείνες, να μπορούν να εξηγήσουν τι πιστεύουν ότι θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα περιφερειακά κέντρα, τις πρωτεύουσε, μιλάω για τη Μάλγα στην Ανταλουσία, για το Λάιτσικ στην ε, Σαξονία, λειψία στη Σαξονία για πόλεις με μεγάλη παράδοση, Πάδοβα για παράδειγμα, ε, δεν ε, είναι περιφερειακές πρωτεύουσες, έχουν όμως και εκείνα άποψη, έχουν πανεπιστήμια και ε, ανθρώπους με άποψη. Θα μπορούσε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει ένα, ένα ρόλο ω προς αυτό. Δεν μιλάμε για την ίδρυση ενός νέου θεσμού, απλώς ένα νέο φόρουμ ε, θέλουμε να δημιουργηθεί. Οποιαδήποτε συζήτηση λαμβάνει χώρα θα έπρεπε να λαμβάνει η χώρα επιτόπου, όχι εδώ, στις πόλεις σε τόπους που μπορούν να έχει πρόσβαση ο κόσμος. Αν γίνει μια συζήτηση λοιπόν στη Μάλαγα, ε, τότε όποιος ε, μένει στη Μάλαγα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν είχε χρόνο να συμμετέχει σε μια συζήτηση ή ότι έγινε μια συζήτηση κάπου που είναι πολύ μακριά για εκείνον να πάει. Είναι πολύ καλύτερο από το να έρχονται ορδές ανθρώπων στις ε, Βρυξέλλες. Βλέποντας το χάρτη της Ευρώπης και βλέποντας το δυναμικό αυτό το δίκτυο, του δικτύου εταίρων ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αν δει κανεί ε, την ε, περιοχή που αφορά χίλιους ανθρώπους, μπορεί να καταλάβει για τι αριθμό πόλεων μιλάμε. Οι μεγάλες πόλεις έχουν δημοτικά συμβούλια, είναι πάρα πολύ καλοί συνομιλητές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν μιλούμε για να ανοίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γραφείο, μιλάμε για συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο, ε, χαμηλού κόστους ε, αλλά υψηλού ωφέλους. Δεν ε, θα έρχεστε σε επαφή μόνο με το Δήμαρχο, με ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο και ολόκληρη την τοπική αρχή θα συνομιλείτε με τα πανεπιστήμια με τα μέσα ενημέρωσης και θα έχετε επιπλέον την ευκαιρία να μιλήσετε με εκλεγμένους ε, εκπροσώπους από ε, πιο απομονωμένες περιοχές, μικρότερες ε, πόλεις, γύρω από τις μεγαλύτερες πόλεις. Νομίζουμε ότι υπάρχει μια υπάρχει τι θέληση για να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα και νομίζω ότι είναι μια ιδέα που έχει νόημα να την αξιοποιήσουμε. Ο στόχος της συζήτηση είναι η Ευρώπη να εξακολουθήσει να αναπτύσσεται ολοκληρωμένα με τη συμμετοχή των πολιτών υποστηριζόμενη από το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας φυσικός σπόνσορας αυτής της διαδικασίας, να μπορεί να θέσει τις ερωτήσεις και να ενθαρρύνει τη διαμόρφωση απόψεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ποιες, ε, ποια θα είναι η αντίδραση των Δήμων ε, και των πόλεων που έχετε, που, σε αυτά που μόλις μας είπατε. Η Άννα Μπόνη τώρα, Άννα Λίσα Μπόνη, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ε, που μας προσκαλέσατε, τη EuroCities, στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική έκθεση πρωτοβουλίας, για μας τουλάχιστον, ε, και πάρα πολύ επίκαιρη ταυτόχρονα. Όπως ακούσαμε, υπάρχουν διάφορες προκλήσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και όλες, όλες συγκεντρώνονται στις πόλεις. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε. Έχω μια σύντομη παρουσίαση, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται στις οθόνες. Μήπως να με βοηθήσει κάποιος. Can somebody help? Can somebody help with... Uh, okay. Oh, anyway. Yeah, it's already... Κάποιος τεχνικός. I've pushed here as I was told. Πατάω τα κουμπιά που μου είπανε, αλλά δεν βλέπω φως. Ah. Okay. So, just a word Έλεγα λοιπόν, να σας ε, συστηθούμε. Τι πρέπει να πατήσω. Τέτοιου είδους πράγματα σκοτώνουν τις ομιλίες πραγματικά. Το βρήκα. Ποιοι είμαστε λοιπόν. Εμείς ε, θεωρούμε ότι είμαστε το δίκτυο στο οποίο απευθύνεται κάποιος για θέματα ε, πόλεων, the go-to network. Πριν από 30 χρόνια αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα οι Δήμοι για να έχουν φωνή οι δήμαρχοι και να συνομιλούν με ε, δικούς τους ε, διάβλους για τα δικά τους προβλήματα. Σήμερα από τους πέντε αρχικούς οι δήμοι αυτοί έχουν γίνει 180 και είναι ένα δίκτυο αναγνωρισμένο που θέλει να επηρεάζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές, να έχει μία φωνή να ε, υπάρχει δικτύωση μεταξύ των μελών και προσπάθεια εξέβρισης λύσεων για τα προβλήματα των πόλων που θα αυξάνουν και την προβολή τους. Σήμερα συμμετέχουν 3.500 πολιτικοί και εμπειρογνώμονες σε αυτή την προσπάθεια. Δεν ξέρω γνωρίζετε το δίκτυο μας γιατί στο Κοινοβούλιο έχουμε συνομιλητή την Επιτροπή Ρέγγι Περιφερειακής Ανάπτυξης και λιγότερο την ΑΦΚΟ, απλώς για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Πάνω από 40 θέματα ε, καλύπτουμε που είναι θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομικά θέματα, ε, κυκλική οικονομία, απόβλητα, κινητικότητα, δημόσια συμβάσεις, ένταξη μεταναστών, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ε, το διαχειρίζονται οι πόλεις. Και πολλά από τα θέματα αυτά είναι και ευρωπαϊκά. Άρα, ως αναγνωρισμένο δίκτυο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, είμαστε σημαντικοί εταίροι και στην, ε, στο αστικό θεματολόγιο. Ακούσατε, είδατε τη μελέτη. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό βήμα αυτό το θεματολόγιο για τις πόλεις. Το αναμένουμε εδώ και 20 χρόνια και κάτι ε, το οποίο κανονικά θα πρέπει να προωθήσει και να βελτιώσει το διάλογο και το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πόλεις αλλά και με τις πόλεις. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που συμμετέχουμε στο σύμφωνο του Άμστερνταμ κλπ. Αλλά παρόλα αυτά Είναι λίγο ευκαιριακή η συμμετοχή των πόλεων και αποσπασματική και θα πρέπει να γίνει πιο συστηματική. Αυτό λοιπόν ήταν το ποιοι είμαστε. Γιατί χρειάζεται ενίσχυση ο ρόλος των πόλεων. Το ακούσαμε και από τους προλαλήσαντες εδώ παρακαθημένους. Ε, δύο-τρία επιχειρήματα. Τα πρώτα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Το δεύτερο σημαντικό στο Ηνωμένο Βασίλειο, α πούμε, με του οποίου συνομιλώ, διαμαρτύρονται σήμερα οι Δήμοι γιατί δεν θεωρούν ότι είναι παρκώς αναγνωρισμένοι στι διαπραγματεύσει για τον Brexit, συγγνώμη, ούτε συμμετέχουν. Και λέει ότι εμεί παράγουμε το περισσότερο ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο, 85%, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και δεν συμμετέχουμε στις συνομιλίες. Όπως σας είπα, σήμερα έχουμε κάποιες ε, δυσλειτουργίες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε στην ομιλία για την κατάσταση στην Ένωση. Μετανάστευση, ανεργία, φτώχεια, κλιματική αλλαγή, όλα αυτά τα θέματα αφορούν τις πόλεις. και στην ομιλία για την κατάσταση στην Ένωση δεν άκουσα ούτε μία φορά τη λέξη πόλη. Είναι σαν να λέμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πραγματικά συγκεντρώνονται στις πόλεις τα προβλήματα στην Ευρώπη και προκλήσεις. Και όχι μόνο αυτό, πάρα πολύ συχνά οι λύσεις είναι επίσης ε, τοπικές. Και προέρχονται από την ίδια την πόλη από διάφορες δυνάμεις, από διαφορετικές προσεγγίσεις. Πολύ συχνά, όταν συγκεντρώνονται όλα αυτά τα προβλήματα σε ένα τόπο, προέρχονται και οι σωστές ε, αποφάσεις από εκεί και οι σωστές λύσεις. Δεν χρειάζεται να είναι πάντα εθνική λύση. Γιατί λοιπόν να ενισχύσουμε το ρόλο των πόλεων, διότι περισσότερο από ποτέ σήμερα υπάρχει μια σαφής ανάγκη σύνδεσης με την τοπική πραγματικότητα. Το 80% της νομοθεσίας εφαρμόζεται στις πόλεις. Θα πρέπει να χτίσουμε γέφυρες ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα ε, της αυτοδιοίκησης ή της διοίκησης. Και το θέμα του, της καλύτερης νομοθεσίας ε, του ευνομοθετή ε, αφορά όλα τα επίπεδα και πολλά από τα προβλήματα και ότι τις δυσκολίες ε, εμφανίζονται σε τοπικό επίπεδο και αυτό δεν το καταλαβαίνουν τα θεσμικά όργανα. Τελικά αν υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα σε ε, αυτό που ζουν οι πολίτες, ποιες είναι οι δυσκολίες τους, τα προβλήματά τους, ε, η καθημερινότητά τους, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει βρει τις λύσεις στο επίπεδο που χρειάζεται. Πρέπει να γεφυρωθεί λοιπόν αυτό το χάσμα. Πώς θα γίνει αυτό μόνο με συνεργασία. Το γιατί λοιπόν είναι σαφές για μας και έχει απαντηθεί. Το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές και είμαι βέβαιη ότι και οι επόμενοι θα το τονίσουν. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε λοιπόν τις σημερινές διευθετήσεις. Όπως σας είπα, περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Εσείς ευρωβουλευτές καθημερινά έχετε επαφή με τους πολίτες και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, σύνδεση με τους πολίτες. Αλλά ταυτόχρονα αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ενισχύσουμε αυτό που λέμε το αστικό θεματολόγιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Urban Agenda. Αυτό ουσιαστικά είναι μια διακυβερνητική ε, διεργασία. Τα κράτη-μέλη έχουν υπογράψει ένα σύμφωνο μεταξύ τους για να δουλέψουν για τα θέματα των πόλεων και ελπίζουμε και με τις πόλεις τις ίδιες. Αυτό βελτιώνεται σιγά-σιγά, αλλά χωράει ακόμα περισσότερη βελτίωση. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακόμα μπορεί να προτείνει και να πιέσει για μεγαλύτερη υποστήριξη, ίσως ένα θεματοφύλακας της πρόοδου. Τι κάνει το Συμβούλιο, το παίρνει αρκετά σοβαρά αυτό υπόψη. Έχουμε δει ότι μετά την Ολλανδική Προεδρία, το επόμενο τρίο δεν προτίθεται να προγραμματίσει ε, συνεδρίαση του Συμβουλίου για θέματα αστικά και για το θεματολόγιο αυτών των πόλεων. Πολύ επικίνδυνο αυτό για μένα. Αν δεν διατηρηθεί ψηλά αυτό το θέμα ε, ε, στην πολιτική, η αστική διάσταση της Ευρώπης δηλαδή, κινδυνεύουμε να χάσουμε μια ευκαιρία να συνδεθούμε με τους πολίτες και να μην απαντήσουμε και λύσουμε τα προβλήματα και της κρίσης. Πολλά είναι εκείνα που μπορούν να γίνουν ε, στην εκπόνηση ε, χάραξη πολιτικών στις πόλεις, το βλέπουμε, ε, στις ομάδες των εμπειρογνωμόνων σπανίως, πάρα πολύ σπάνια συμμετέχουν πόλεις. Στην Επιτροπή Περιφερειών αρχίζουν να κάνουν μελέτες αντικτύπου ε, στο αστικό περιβάλλον, δειλά-δειλά, αλλά και πάλι χωράει εκεί βελτίωση. Και όχι να παίρνει τηλέφωνο πέντε λεπτά πριν, άμε πώς να φέρετε πέντε ή δέκα εμπειρογνώμονες από πόλεις να κοιτάξουν αυτή την οδηγία. Επίση χρειάζεται συντονισμό πολιτικής μεταξύ Γενικών Διευθύνσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό μεν βελτιώνεται, αλλά θα μπορούσε να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω. Και πώς μπορούμε να έχουμε ανοιχτή ατζέντα με 12 ομάδες εργασίας. Δεν ξέρω αν... Ε, γνωρίζετε πώς λειτουργεί, αλλά είναι διάφορες ομάδες με διάφορους εμπειρογνώμονες. Όλα αυτά πώς μπορούν να ενταχθούν στην, ε, ε, στο ΡΕΦΙΤ για καλύτερη νομοθεσία. Ο κόσμος εργάζεται, δαπανά πόρους, χρόνο, όλα αυτά είναι θελοντικά και όλα αυτά μένουν στα συρτάρια ή σε ράφια και δεν ε, εντάσσονται ή δεν έχουν επιρροή στον κύκλο λήψη αποφάσεων και πολιτικών. Αυτό θέλω να το τονίζω. Δεν είπα ότι δεν χρειάζεται το αστικό θεματολόγιο. Πραγματικά εμείς δίνουμε και το αίμα μας για να ε, προχωρήσει αυτή η προσπάθεια και να ευοδοθεί. Αλλά μπορεί να ενισχυθεί το κοινοβούλιο, μπορεί να παίξει ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε κάποιους βουλευτές που ενδιαφέρονται και προωθούν τα θέματα, αλλά δεν νομίζω. Νομίζω ότι στις περισσότερες επιτροπές δεν κυριαρχεί αυτό το θέμα των πόλων. Και τελειώνω. Ο στόχος είναι κοινό για όλους. Να προωθήσουμε μια Ευρώπη που να έχει νόημα για τους πολίτες μας. Η διαφάνεια δεν έρχεται, αλλά θα σας τα πω εγώ. Να προωθήσουμε λοιπόν μια Ευρώπη που να έχει νόημα για τους πολίτες, γιατί πραγματικά δεν έχει να συνεχίζουμε αυτή την αναντιστοιχία. Και ως ε, Eurocities το δίκτυό μας έχει δεσμευτεί με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Έχουμε κινήσει μια εκστρατεία που λέγεται η Ευρώπη για τις πόλεις και πόλεις για τους πολίτες. Καλύπτουμε 130 εκατομμύρια κατοίκων βασικά και δίνουμε φωνή στους πολίτες για να εμπνεύσουν τη συζήτηση για την Ευρώπη. Τι θέλω αυτή την τελευταία διαφάνεια που δεν κατεβαίνει, μάλιστα, γιατί το μήνυμα που σας απευθύνουμε είναι συνεργαστείτε μαζί μας, γιατί μόνο από κοινού μπορούμε να προχωρήσουμε και να έχουμε ένα πιο θετικό αφήγημα για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Very Ευχαριστώ. Λουκμάν, Μάτες, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επόλεων και Περιφερειών και και σύμβουλος, ε, δημοτικός σύμβουλος στο Ρεζελάρ να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε ε, για την ε, πρωτοβουλία σας. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασχολούνται με την υπόθεση των πόλων και ιδιαίτερα τους παρόντες. Γιατί καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι οι, ότι οι βουλευτές ε, έχουν φυγαδευτεί κάπου στις χώρες τους και ψάχνουν την πόλη τους. Ακούω τους συναδέλφους και ε, διαπιστώνω ότι έχουμε πολλά κοινά και μεγάλη συναντήληψη. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και μεγάλες διαφορές ήδη στη χρήση της ορολογίας που χρησιμοποιούμε. Όταν λέμε περιφέρειες, τι εννοούμε. Όταν λέμε πόλεις, τι εννοούμε. Μιλάμε για τα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα, τα μεγάλα αστικά κέντρα της μεγάλου πόλης όλες τις μικρότερες, γιατί υπάρχουν ε, και πόλεις που δεν είναι πολύ μεγάλες αλλά είναι σημαντικές. Και κάπου οξύνονται τα προβλήματα σε ε, μεγαλύτερη κλίμακα, αλλά δεν είναι αναγκαστικά αυτή η πραγματικότητα. Λοιπόν, ε, συμφωνούμε γενικά και σε αυτά που είπε η ο εκπρόσωπος της Επιτροπής των Περιφερειών αισθάνομαι ότι ο Πρόεδρος και όλη η Επιτροπή των Περιφέρειών έχει πολύ μεγάλη ε, εικόνα και αντίληψη για το τι κάνει η τοπική ε, αυτοδιοίκηση. Ο Λάμπερτς ο ίδιος, ο πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, διατέλεσε και δήμαρχος. Τι είναι το CMR, ε, πάρα πολύ γρήγορα. Από την αρχή είναι μια οργάνωση ε, που έχει καταβάλει προσπάθειες ε, να υλοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση από την ιστορία, από την καταβολή ε, από την ΕΚΑΧ και λοιπά ήδη από το 1951 50 δήμαρχοι από τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τους κάτω χώρες το Λουξεμβούργο, ακόμα και την ε, Ελβετία, είπαμε ότι θα κάνουμε ένα τέτοιο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να υποστηρίξουμε μια Ευρώπη ειρηνική, ενωμένη, ευημερούσα και ε, από τότε έκαναμε αυτή την προσπάθεια. Και σήμερα είμαστε ε, μια οργάνωση φόρουμ ε, μια ομπρέλα όπως τη λέμε για 60 διαφορετικές ε, οργανώσεις και ενώσεις τις οποίες συγκεντρώνουμε σε 42 χώρες παρακαλώ. Σε κάποιες χώρες έχουμε 2-3, σε 7 χώρες έχουμε μία ε, μεγάλη οργάνωση, κεντρική ένωση δήμων και κοινοτήτων, σύνολο 130.000, 130.000 φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για ε, λόγους συμβουλευτικούς. Άρα έχουμε αποδείξει και την πίστη μας και την αφοσίωσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές φορές συμμετέχουμε σε συζητήσεις ας πούμε για τη συνθήκη της Λισαβόνας ή και Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 και τα λοιπά. Ή ε, όταν συζητάμε για πολιτική συνοχής, για στρατηγικές συνοχές. Αλλά ο ρόλος μας είναι ακόμα υποβαθμισμένος ή περιορισμένος. Η οταν συζηταμε για πολιτικη συνοχή για στρατηγικες συνοχες αλλα ο αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή κανονικά είναι ο τόπος όπου ο κόσμος ζει τα προβλήματα και εκεί ε, πρέπει να λύνονται. Είτε πρόκειται για το κλίμα, είτε πρόκειται για την κινητικότητα, για τα νητρικά και την ρήπανση του εδάφους. Εκεί είναι η πίεση της πολιτικής. Ε, εκεί αισθάνεται την πίεση η τοπική αυτοδιοίκηση και εκεί ακόμα ο πολίτης εμπιστεύεται πολύ ε, τους ηθήνοντες και τους ε, τοπικούς άρχοντες. Και εκεί η Ευρώπη ε, μπορεί να αποδειχθεί. Ένας Ινδός έχει γράψει πρόσφατα ένα βιβλίο The Age of Anger, ε, η εποχή του, of anger μάλλον, η εποχή του, του θυμού, ε, γιατί δείχνει ότι ε, ο κόσμος έχει εξοργιστεί, έχει θυμώσει και ψάχνει από διοπομπαίους τράγους στην κεντρική πολιτιστική σκηνή και πολλές φορές η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας μεσολαβητής το 75% το 80% της νομοθεσίας εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν και το Συμβούλιο μας των Δήμων και Κοινοτήτων ε, χρειάζεται μια συμμαχία ε, σε τοπικό επίπεδο. Αν το δούμε ιεραρχικά, ε, Νομίζω έχουν παρέρθει οι καιροί όπου υπήρχε η ιεραρχία αυτή η κάθετη, όπου υπάρχει ένα στρώμα διοίκηση πάνω από το επόμενο. Όλο και περισσότερο ε, ε, έχουμε οριζόντια ε, διάρθρωση, ο καθένας σέβεται τις αρμοδιότητες του άλλου, δεν υπάρχει κάθετη οργάνωση και έτσι υπάρχει καλύτερη συνεργασία. Και τι μαθαίνουμε λοιπόν, ότι θα πρέπει να μας αφορά και να συμμετέχουμε σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα στάδια. Από την αρχή, από τη σύλληψη, τη στρατηγική, την ε, ε, κατάρτιση, την υλοποίηση, ακόμα και την εκτίμηση και την αξιολόγηση. Θα πρέπει να είμαστε παρόντες το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών. Γιατί καλύτερα ξέρει η τοπική αυτοδιοίκηση πώς εφαρμόζονται όλα αυτά επί τόπου και πώς λύνονται τα προβλήματα. Ακόμα και το κόστος μειώνεται, αν το δούμε, με πρωτοβουλίες ε, να είναι λιγότερο το πλαίσιο το ρυθμιστικό, το γραφειοκρατικό ε, και να έχουμε λύσεις ε, που να λειτουργούν στην πράξη και όχι απλώς στα χαρτιά. Άρα Τι λέει λοιπόν το CMR, ε, το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών. Μην το παρακάνετε στις λεπτομέρειες, αφήστε μας ένα περιθώριο ελιγμών. Κάθε πόλη, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει την ιστορία της, ε, έχει ένα παρελθόν. Στη Φλάνδρα ας πούμε. Δεν έχουμε μεγάλες πόλεις. Και η η πόλη των Βρυξελών δεν είναι μεγάλη πόλη. 100.000 κατοίκους έχει το πολύ πολύ ο Δήμος των Βρυξελών δεν μιλώ για την περιφέρεια. Τρία επί τρία χιλιόμετρα είναι η πόλη των Βρυξελών. Σιγά τη μεγαλούπολη. Άρα πρέπει να καταλαβαίνουμε ε, τη διάσταση αυτή την τοπική ε, και στην Ευρώπη να έχουμε την αρχή της επικουρικότητας και να την εφαρμόζουμε. Και την οικονομική ε, οικονομική αυτονομία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης το λέει να υπάρχει αυτονομία οικονομική για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό απέχει πόρο από την πραγματικότητα. Ε, πολλές αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης εξαρτώνται από τη φορολογική κυριαρχία ε, των κρατών μελών και δεν μπορούν να απτύξουν ένα στρατηγικό όραμα ούτε να δουλέψουν σωστά. Ε, διαχείριση, διακυβέρνηση και εταιρική σχέση να είναι ευρύτερη η διοίκηση, πέρα από την πολιτική και μόνο συμμετέχει και η κοινωνία και όλα τα επίπεδα πολιτικής. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η εταιρική σχέση, το partnership. Έχουμε καλές εμπειρίες, ε, υπάρχουν ενδιαφέρουσες μελέτες και στη δική μας οργάνωση και ε, έχουμε την βελγική εμπειρία αλλά και άλλων κρατών μελών και ενθαρρύνω και τον εισηγητή και τους εμπειρογνώμονες να ανατρέξουν σε αυτές τις μελέτες και τις εκθέσεις και να τα συμπεριλάβουν στην έκθεση. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν ε, εργαλεία και δομές πιο προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα και ε, να αλλάξουν και οι νοοτροπίες και οι συμπεριφορές. Καταλαβαίνουμε ότι από τη μια χρειάζεται ε, μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω μέχρι ένα συγκεκριμένο επίπεδο αλλά εξευρεθεί και εκείνη η ισορροπία που χρειάζεται για να λαμβάνονται καλύτερα οι αποφάσεις. Και στο βαθμό που θα γίνουν αυτά θα υπάρχει ένας διάλογος και όχι απαξ, όχι να, επειδή το ζητάει κάποιος ή επειδή έγινε ένα επεισόδιο, αλλά επειδή το θεωρούμε σημαντικό και ε, ε, παίρνουμε σοβαρά υπόψη και το συνομιλητή μας, τότε θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Να έχουμε ένα διάλογο ε, με κριτικό πνεύμα, με ειλικρίνεια και αμεσότητα, αλλά με εταίρους που μπορούν να είναι ένας πολλαπλασιαστής, ένας ενισχυτής, ένας επιταχυντής σωματιδίων μάλιστα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όλες τις γενιές και τις επερχόμενες. Ευχαριστώ. Ο Γιάνν Όλμπριχτ ε, θα πάρει το λόγο. Όπως είπα και στην αρχή, ο κ. Σουγιαντόφσκι... Ε, συμμετέχει ισότιμα δυνάμει του άρθρου 54 ε, με τον κύριο Όλμπριχτ σε αυτό το θέμα. Παρακαλώ, ξέρετε τους κανόνες, ε, σεβαστείτε τους, βεβαίως. Μια και ο εισηγητής είναι Πολωνός, θα μπορούσα να μιλήσω πολωνικά, αλλά για να με καταλάβουν οι φίλοι από τις πόλεις που θα μπορούσα τελικά να μιλήσω αγγλικά. Το βασικό θέμα είναι είναι πια είναι η θέση των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο μας. Αναγνωρίζεται ο ρόλος τους στο ευρωπαϊκό σύστημα ή όχι. Θα σας πω ποια είναι η άποψη της Επιτροπής, ε, των Περιφερ... Ε, της ε, Επιτροπής του Κοινοβουλίου. Εμείς θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της περιφερειακής πολιτικής. Έχουμε δύο διαδικασίες στην Ευρώπη. Η μία είναι η περιφερειοποίηση, που είναι μια διοικητική διαδικασία. Αφορά τις αρμοδιότητες των περιφερειών, το ρόλο, το ρόλο τους στο συνταγματικό πλαίσιο ε, των κρατών μελών. Η περιφερειοποίηση είναι ε, η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των πόλεων. Η επικουρικότητα όμως είναι ότι δεν πρέπει να αγγίξουμε τις πόλεις ε, και ποιο είναι ο ρόλο του στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο των κρατών μελών. Ε, η περιφερειακή πολιτική είναι η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορά τι περιφέρειες έτσι, των ΝΑΤΣ 2 και είναι ευρωπαϊκό θέμα, ευρωπαϊκή υπόθεση. Ε, οι περιφέρειε τελικά είναι ευρωπαϊκό θέμα ή όχι από τη σκοπιά τη περιφερειοποίηση, ε, διοικητικά και νομικά, όχι. Είναι θέμα επικουρικότητα. Κανένα στι Βρυξέλλε δεν αποφασίζει για τι περιφέρειε. Αντίθετα, τα λεφτά τα οποία πηγαίνουν στι περιφέρειε, ε, γι' αυτό έχουμε την περιφερειακή πολιτική. Έχουμε ακριβώ την ίδια κατάσταση με τι πόλει. Και όμω δεν τη συζητάμε καθόλου τι πόλει. Με βάση την αρχή τη επικουρικότητα, η δομή του συγκεκριμένου κρατου μέλους του Ηνωμένου Βασιλείου, ας πούμε, το οποίο έχει μια πολύ ειδική, έχουν μια ειδική μάλλον θέση οι πόλεις. Ε, η αρμοδιότητα αυτή είναι βρετανική αρμοδιότητα. Ε, μπορούν να αποφασίσουν αν θέλουν μικρές, μεσαίες, μικροπολιτικέ ε, μικροπολιτικές πόλεις, τα κράτη-μέλη αποφασίζουν. Κανένας δεν μπορεί να παρισφρήσει αυτό. Από την άλλη, τα λεφτά, τα ευρωπαϊκά λεφτά που πηγαίνουν ε, στις πόλεις περνάνε μέσα από τις περιφέρειες. Όλο και περισσότερο τώρα προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε οι πόλεις μάλλον να είναι απευθείας δικαιούχοι ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τελικά θέλουμε να ανακατευθούμε τις πόλεις ή όχι. Μερικές φορές ε, επικαλούμαστε την αρχή της επικουρικότητας για να μην το κάνουμε. Πριν από χρόνια ε, συζητούσαμε εδώ, πέρα για να, συζη... να αναπτύξουμε μία αστική πολιτική για τις πόλεις. Να μην μειώσουμε την αρχή της επικουρικότητας και τη σημασία της, αλλά να ενισχύσουμε το ρόλο των πόλεων, να αναγνωρίσουμε το ρόλο των πόλεων στο σύστημα. Οι πόλεις πρέπει να έχουν λόγο. Οι τοπικές αρχές βεβαίως να έχουν λόγο οι φορείς των πόλεων θα πρέπει να έχουν λόγο. Γι' αυτό το σύμφωνο του Άμστερνταμ ε, έλεγε αυτά που έλεγε για τις πόλεις και δεν συμφωνώ με τον εισηγητή. Η κατάσταση είναι πειραματική εκεί. Ήταν πειραματική μάλλον εκεί στο σύμφωνο του Άμστερνταμ. Τώρα για πρώτη φορά να γνωρίσουμε το ρόλο των πόλεων στο σύστημα. Θυμάμαι όταν η κυρία Χιούμπνερ ήταν επίτροπος συζητούσαμε το ρόλο τότε των ε, διαχειριστικών αρχών των κρατών μελών. Τώρα έχουμε εταιρικέ σχέσεις και για πρώτη φορά οι πόλεις κάθονται σε, ένα, σε μια στρογγυλή τράπεζα όπου όλοι συζητάνε ισότιμα. Μαζί με το, τους επιτρόπους, μαζί με τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων και οι εκπρόσωποι των πόλεων. Και είναι δύσκολο πείραμα, ειδικά για την Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, να αντιμετωπίσουν σαν ισότιμους τους εκπροσώπους των πόλεων και να συζητήσουν τα πραγματικά προβλήματα. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το follow-up. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή ε, να μιλήσουμε όλοι για τις πόλεις. Έξι επίτροποι ε, ασχολούνται με αυτό το θέμα. Είναι συναρμόδιοι για το θέμα των πόλεων. Το θέμα είναι πώς θα ε, αναγνωριστεί επίσημα στο σύστημα ο ρόλος των πόλεων. Των πόλεων. Η περιφερειοποίηση είναι θέμα επικουρικότητας. Από την άλλη, τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορεί να επηρεάσουν την ε, διαδικασία της ε, περιφερειοποίησης. Τα ευρωπαϊκά λεφτά μπορούν να ενισχύσουν τις περιφέρειες ή να μειώσουν τις περιφέρειες. Η περιφερειακή πολιτική στέλνει λεφτά στις πόλεις, αλλά ενισχύει τις πόλεις ή μειώνει τη σημασία των πόλεων. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα παράλληλα. Εμείς στη Ρέτζι θα γνωμοδοτήσουμε και θα πούμε ότι αυτή είναι η στιγμή όχι να μιλήσουμε για τις πόλεις, αλλά για να κάνουμε κάτι και να γνωρίσουμε το ρόλο του στο σύστημα. Να αλλάξουμε το σύστημα, να γνωρίσουμε τις πόλεις στο σύστημα και να ορίσουμε πολύ σωστά ποια είναι η θέση τους. ξεκινήσαμε την όλη διαδικασία με τη χάρτα της λειψείας. Καλά είναι, καλό είναι να συνεχίσουμε. Ε, στο κήτο του Εκουαδόρ κάναμε μία συνάντηση όπου ο ΙΕ... Ε, ασχολούνταν με το στόχο της χιλιετίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, παριθμό 11. Ποιο ήταν το βασικό πρόβλημα στον ΟΗΕ επί μήνες. Οι περισσότερες χώρες, κυρίως οι αφρικανικές και οι ασιατικές, δεν ήθελαν να μπει στο κείμενο η λέξη πόλης. Θέλαν τις πόλεις, ναι, αλλά σαν συνοθήλευμα. Όχι τις τοπικές αρχές, όχι τους τοπικούς φορείς, γιατί ξέρανε ότι η πόλη είναι στα χέρια των κυβερνήσεων. Και χρειάστηκαν μήνες για να μπει μία λέξη στο κείμενο και να λέμε ότι στα, στα πλαίσια του νέου θεματολογίου για τα αστικά θέματα θα πρέπει να αναγνωριστούν οι πόλεις. Αυτό σας το λέω έτσι είναι ήδη παραδείγματος. Το θέμα είναι ενδιαφέρον και όπως και το Brexit και και εδώ για το θέμα των πόλεων έχουμε την κατάλληλη ευκαιρία για να κάνουμε κάτι. Ας αναγνωρίσετε και εσείς στην Επιτροπή σας το ρόλο των πόλεων. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί στο όλο σύστημα η θέση των πόλεων. Ο κύριος Χαουρέγγι. Θέλω και εγώ να συνεισφέρω στον προβληματισμό που μόλις έκανε ο συνάδελφος. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ουγιαρντόφσκι για την πρωτοβουλία αυτή να βάλει στη συζήτηση το θέμα των πόλεων. Στη συζήτηση της ΑΦΚΟ εννοώ. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο, πολύ σωστό και ιδίω μετά τις παρεμβάσεις των συναδέλφων θεωρώ ότι είναι σωστό. Ε, μιλάω εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Και θα ήθελα να σας πω ότι εμείς οι σοσιαλιστές συμφωνούμε με τον εκπρόσωπο του Λαϊκού Κόμματος ως προς την ιδέα ότι η πόλεις αποτελούν τμήμα του θεσμικού, ας πούμε, πλαισίου μας. Έτσι καταλαβαίνουμε και την ευρωπαϊκή θαγένεια μέσω των πόλεων έτσι, και τη σημασία τους. Και νομίζω ότι οι συνεισφορές των εμπειρογνωμών είναι πολύ σημαντικές. Τους ευχαριστώ. Και μας μιλάνε για αυτή την ιδέα ότι δεν υπάρχει σήμερα ιδέα της δημοκρατίας εάν δεν υπάρχει έντονη συμμετοχή των πόλεων, των πολιτών μέσα από τις ε, πόλεις τους, έτσι, στις πόλεις οποίες ανήκουν και προέρχονται. Εμείς φτιάξαμε μία ε, έκθεση για την ηλεκτρονική δημοκρατία, δηλαδή τις δυνατότητες που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας. Και το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να φέρουμε τη δημοκρατία στις ε, πόλεις, μέσα από τις διαβουλεύσεις, μέσα από την χρήση των νέων τεχνολογιών, ούτω ώστε οι πολίτες να συμμετέχουν πιο άμεσα σε θέματα, ε, απλούστερα, να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Δεν μιλάω για δημοψηφίσματα που καθορίζουν ταυτότητά μας, αλλά μιλάω για πιο καθημερινά πράγματα. Μέσα λοιπόν από αυτέ τι νέες τεχνολογίες ε, ε, έχουμε τεράστιες ευκαιρίες για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία. Αυτά που υπόθηκαν για την ε, ενίσχυση των τοπικών πολιτικών, για την ε, διάδοση των καλύτερων πρακτικών, για τη διάδοση των γνώσεων κτλ. Όλα αυτά νομίζω δείχνουν τη σημασία των πόλεων. Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις που αντιτίθενται όμως αυτή την ιδέα της συμμετοχής των πόλεων. Καταρχάς, υπάρχει μια ανομοιογένεια ε, των ε, τοπικών αρχών. Εμείς έχουμε 8.000 δήμους και κοινότητες. Και έχουμε τεράστιες διαφορές. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ μεγάλους δήμους και πάρα πολύ μικρές κοινότητες. Από την άλλη. Είδα την έκθεση που ετοίμασε το Κοινοβούλιο. Και βλέπω τα ποσοστά εκπροσώπησης και τα λοιπά. Τα ποσά, την εκπροσώπηση μάλλον. Λόγω της διαφορετικότητας αυτής θα πρέπει την ε, τοπική αυτή εκπροσώπηση να την ε, συνδέσουμε ε, με τον αριθμό των πολιτών. Η Ευρώπη επίσης ε, μπορεί να μας βάλει πολλά εμπόδια γραφειοκρατικά. Με αυτόν τον τρόπο μας κατακρίνουν οι πολίτες γιατί είμαστε υπερβολικά γραφειοκρατικοί και δεν είμαστε αποτελεσματικοί. Επίσης το τρίτο πρόβλημα είναι ότι οι αποφάσεις για οι πολιτικές αποφάσεις ας πούμε εξαρτώνται από τις χώρες. Ε, κάθε χώρα έχει τους δικούς, τις, και στις κανόνες και αποφασίζουν πώς θα μοιράσουν την εξουσία, έτσι, ανάλογα με τις παραδόσεις κτλ. Τελειώνω. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ τον Πολωνό εισηγητή και θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι πάμε προς, ε, μια, ένα, προς ένα ομοσπονδιακό σύστημα. Και δεν θέλω να δημιουργήσω δυσαρέσκεια σε κανένα. Ε, υπάρχει ε, μια τάση οργάνωση της δημοκρατίας μέσα από τους δημόσιους αυτούς χώρους. Έτσι. Έχουμε την περιφέρεια, τις αυτόνομες κοινότητες, τα lender, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσετε. Αυτό είναι. Και από την άλλη, το κράτος, ε, τα κράτη-έθνη ας πούμε και την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε την ταυτότητα, έχουμε την επικουρικότητα, έχουμε την αλληλεγγύη και την αποτελεσματικότητα. Αυτές είναι τέσσερις αρχές. Και με βάση αυτό το σχήμα, ας πούμε, νομίζω ότι είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τη θέση των πόλεων προς το συμφέρον της δημοκρατίας μας. Ευχαριστώ, Ραμόν. Τελειώσαμε τη συζήτηση. Αν θέλει κανείς να απαντήσει στα σχόλια της ερωτήση, μπορώ να σας δώσω ένα λεπτό, γιατί έχουμε πάρα πολύ καθυστερήσει. Sorry, nobody wants to speak. Uh, so you are working against your interests now, you know. Θέλει να πάρει το λόγο. Ναι, αλλά είναι η επόμενη έκθεση δική σου και αν μιλήσεις πάρα πολύ τώρα θα είναι εναντίον σου γιατί μπορεί να αναβληθεί επόμενη, το επόμενο θέμα. Απλώς να πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει τώρα αυτή η αναστάτωση με το ζήτημα της ε, Καταλωνίας ε, και επίσης έχουμε πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σε ολόκληρη την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ανατολή και στη Δύση. Γι' αυτό το λόγο, εγώ πιστεύω ότι αυτό το ζήτημα των πόλεων είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν εστιαστούμε στην Ευρώπη των πόλεων, υποκαθιστώντας την παλιά ιδέα της Ευρώπης των περιφερειών, μπορεί να ε, μπορέσουμε να επιλύσουμε και να αντιμετωπίσουμε επιτυχέστερα τις προκλήσεις αυτές που μόνο θα αυξηθούν ε, κατά τα επόμενα έτη. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια πολύ σημαντική πολιτική στρατηγική γιατί μερικές φορές ε, η Ευρώπη των περιφερειών ε, είχε αποτελέσει το αίτιο τέτοιου είδους ε, αναταράξεων. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θέλει κανείς ένα λεπτό να πει οτιδήποτε. Αν όχι, τότε να δώσω το λόγο στον ε, εισηγητή για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ε, εμπειρογνώμονες για τις παρουσιάσεις τους, για τις εξαιρετικές τους προτάσεις. Να ευχαριστήσω επίσης ε, και τους ε, ευρωβουλευτές για τις παρεμβάσεις τους εγώ νομίζω ότι είναι, έχει πια έρθει η χρονική στιγμή να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε τις πόλεις στο, στη θεσμική αρχιτεκτονική της Ένωσης και υπάρχουν πολλοί λόγοι για να γίνει κάτι τέτοιο, κυρίως δύο που αναφέρθηκαν σήμερα. ο σημαντικότερος ρόλος των ε, πόλεων στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανάγκη ε, αξιοποίησης, ενθάρρυνσης του δυναμικού που υπάρχει, όπως είπε και ο καθηγητής Ματίγια. Ε, δεν θα ήθελα να υπάρξει παρανόηση. Το σύμφωνο του Άμστερνταμ και η σχετική πλατφόρμα είναι πολύ καλά. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να υποτιμήσω τη σημασία τους. Πιστεύω απλώς ότι έχει επιτέλους έρθει η στιγμή να ε, ξαναδούμε σοβαρά και να ενισχύσουμε τη θέση των πόλεων γιατί έτσι βασιζόμαστε στην ε, ε, συνεργασία μεταξύ των πόλεων. Εγώ δεν θέλω να αλλάξω κάτι που υπάρχει με κάτι διαφορετικό. Ε, είναι ένα κοινό ζήτημα της Επιτροπής Ρέτζη και ε, της δικής μας ε, Επιτροπής. Ναι, αλλά θα θέλαμε να κλείσουμε αυτό το ε, σημείο της ημερήσιας διάταξης και θα θέλαμε να σας ζητήσουμε δεν, δεν χρειαζόμαστε ε, χρονοδιάγραμμα. Ποιες είναι οι ημερομηνίες που μπορούμε να περιμένουμε. Δεν είστε βέβαιος από ό,τι κατάλαβα για το χρονοδιάγραμμα αυτό. Δύο μήνες θα έλεγα για το σχέδιο έκθεσης. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα νομίζω και δεν είναι πάνω από δύο μήνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με βέβαια ότι δεν είναι η τελευταία φορά που συναντιόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις, ε, τη συμβολή σας, όλους τους προσκεκλημένους. Μεταδίδεται και στο διαδίκτυο η συνεδρίαση από την αρχή. Οπότε ό,τι είπατε δεν ε, παραμένει μόνο σε αυτή την αίθουσα. Παύλο Ράντζελ τώρα, έκθεση ε, ιδίας πρωτοβουλίας για την εφαρμογή των διατάξεων συνθήκης ε, σε σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια. Σήμερα θα γίνει η παρουσίαση της μελέτης ε, που εκπώνησε η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το EPRS. Να μας κάνετε εσείς μια εισαγωγή και μετά θα ακούσουμε τον Μίλαν Ρέματς ο Ράντζελ. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε απευθείας στην παρουσίαση τη έκθεση και μετά θα κάνω μερικά σχόλια για το έγγραφο εργασία που έχω προετοιμάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μίλαν Ρέματ λοιπόν να μα παρουσιάσει την ε, εκ των υστέρων αξιολόγηση της υπηρεσίας ε, ε, έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω πέντε λεπτά, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας υποβάλλατε αυτό το έγγραφο εργασίας. Εμάς ε, μας ζητήθηκε Μιλάμε για το τμήμα C ε, των, των, της εκ των αξιολόγησης. Ε, μας ζητήθηκε να εκπονήσουμε δύο έγγραφα, μία ε, μελέτη σε σχέση με την ε, συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια για ζητήματα της Ένωσης και ένα ακόμη ε, έγγραφο. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μία ανάλυση από την έρευνα που κάναμε ε, για τη θέση των ε, οργάνων της Ένωσης. Δυστυχώς κλείνει το μικρόφωνο του μιλητή. Έγινε επίσης και μία έρευνα μεταξύ των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο. Υπήρξε μία έρευνα και μία ε, μελέτη που δημοσιεύθηκαν προσφάτως και φαντάζομαι ότι υπάρχουν στον ηλεκτρονικό σας φάκελο. Ποιος ήταν ε, ο στόχος τώρα του εγγράφου μας ήταν ουσιαστικά να υπάρξουν συνοδευτικά έγγραφα ε, προς το έγγραφο του εισηγητή και να υπάρξουν και κάποιες πληροφορίες ε, ως ιστορικό ε, για την έκθεση του. Υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα τα οποία έχουν εκπονηθεί εντός και εκτός υπηρεσίας μας. Έχουμε προσπαθήσει εμείς να κάνουμε μία επισκόπηση των εφισταμένων δεδομένων. Η μεθοδολογία μας λοιπόν βασίστηκε σε έρευνα που έγινε ε, από την υπηρεσία μας αλλά και σε εμπειρική έρευνα. Δεν ε, μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε βέβαια όλα ε, τα στοιχεία. Συμπεριλαμβάνονται πάντως όλα τα έγγραφα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Κοινοβούλιο, από το Συμβούλιο και υπάρχουν κάποια τμήματα που αφορούν την ΚΟΖΑΚ που είναι η διάσκεψη των κοινοβουλίων ε, για τα ε, ζητήματα της Ένωσης, όπως επίσης και η διάσκεψη των προέδρων των κοινοβουλίων. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε μια επισκόπηση και ανάλυση όλων αυτών των ε, δημοσίως διαθέσιμων ε, πηγών. Έγινε και μια έρευνα μεταξύ των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων που ήταν ανώνυμοι. Έγινε τον ε, Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2017. Εμείς ζητήσαμε από τους εθνικούς εκπροσώπους να μας απαντήσουν σε 11 ερωτήσεις και λάβαμε ε, περίπου 90% ε, από 90% λάβαμε απαντήσεις και μας έκαναν μάλιστα και κάποια σχόλια σε σχέση με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την διοικητική πλευρά της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, βασικά πορίσματα λοιπόν της μελέτης μας είναι τα εξής. Α, δουλεύει τώρα και η τεχνολογία. Πάλι δεν δουλεύει. Uh, with regards to the main results of the study. Λοιπόν, τα βασικά ε, πορίσματα της ε, μελέτης μας είναι ότι από το 2007 από τότε δηλαδή άρχισε να υπάρξει μια ενίσχυση της ε, συμμετοχής των Εθνικών Κοινοβουλίων, η οποία όμως παραμένει περιορισμένη και παραμένει περιορισμένη ε, στο μηχανισμό έγκαιρης προεδοποίησης και τη διακοινοβουλευτική ε, συνεργασία. Επίσης, οι αιτιολογημένες γνώμες του Εθνικού Κοινοβουλίου μερικές φορές δεν μπορούμε να ξέρουμε αν όντω καθυστερεί ή έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση μιας διαδικασίας ε, υπάρχει περίπτωση λοιπόν να ενισχύεται η θέση των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, στα ενωσιακά ζητήματα, αυτό ήταν το συμπέρασμα, και επίσης έχουμε δει ε, μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίων. Λοιπόν, Ως προς τα αποτελέσματα τώρα της μελέτης, της, συγγνώμη, της έρευνας, είδαμε ότι υπήρξε μια γενική ικανοποίηση των εκπροσώπων Εθνικών Κοινοβουλίων με τη θέση ε, και την παρουσία τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμως έθεσαν πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προσέγγιση και την πολιτική πληροφόρηση από, το Κοινοβούλιο, από την Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των πολιτικών ομάδων και ειδικότερα από τις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τρίτο κύριο πόρισμα είναι ότι το υφιστάμενο δίκτυο των εκπροσώπων Εθνικών Κοινοβουλίων θεωρεί ότι όντως ενισχύθηκε η συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλίων και επίσης η παρουσία των εκπροσώπων εθνικών κοινοβουλίων ουσιαστικά ε, δίνει περισσότερες δυνατότητες ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Ωραία. Να σας δείξω απλώς την ικανοποίηση των ε, ε, εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, σε σχέση με την ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περίπου 53% των εκπροσώπων είναι ικανοποιημένοι με την πολιτική του, της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 59% εξ αυτών είναι ικανοποιημένοι με την πολιτική ενημέρωση των πολιτικών ομάδων. Υπήρξε μία έλλειψη ικανοποίησης ε, όσον αφορά την ε, ενημέρωση από τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οργάνωση των ε, συνεδριάσεων του των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων ε, είχε παρουσιάσει προβλήματα κατά την άποψη των εκπροσώπων. Αυτά ήταν τα ε, βασικά ε, αποτελέσματα της μελέτης μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στον Παύλο. Ευχαριστώ πολύ. I'll start to thank to... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την η υπηρεσία EPRS και ιδιαίτερα τον κύριο Ρεμάκ διότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η δουλειά που έκαναν η μελέτη και όπως έχουμε ακούσει και προηγουμένως ε, ε, υπήρξε εκτενέστατη ανταλλαγή απόψεων και πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο αυτό για την υπηρεσία. Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και πάρα πολύ ειλικρινής. Έχετε το έγγραφο εργασίας το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα, αυτά τα θέματα καλύτερα σε προηγούμενη συνεδρίαση με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων, οπότε θα έρθω κατευθείαν στα συμπεράσματα, τα βασικότερα. Το πρώτο που θα πρέπει πάντα να τονίζουμε και να υπογραμμίζουμε είναι ότι ο βασικός θεσμικός και συνταγματικός ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των ίδιων των κυβερνήσεών τους. Έχουν εργαλεία ισχυρά και μέσα να εκφράσουν και να διαμορφώσουν τη θέση του κράτους τους στα Συμβούλια Υπουργών, ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και αυτό παραμένει βασική συνταγματική εξουσία που έχουν τα Εθνικά Κοινοβούλια στην ισορροπία των εξουσιών ε, στο ευρωπαϊκό θεσμικό και συνταγματικό οικοδόμημα. Από εκεί και πέρα ελέγχουν την επικουρικότητα τα κοινοβούλια. Πιστεύω ότι τους αρέσει η ιδέα αυτών των ε, ε, πορτοκαλί κίτρινων καρτών, αλλά είναι λίγο δυσαρεστημένοι με την εμπειρία της κίτρινης κάρτας και το μηχανισμό της έγκαιρης προειδοποίησης. Για ποιο λόγο? διότι είναι πεπισμένα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερμηνεύει πάρα πολύ αυστηρά την αρχή της επικουρικότητας και περιοριστικά. Και πρέπει να σας πω ως νομικός και εμπειρογνώμων περί τα συνταγματικά θέματα ότι ακόμα και οι δικές μας νομικές υπηρεσίες έχουν πάρα πολύ αυστηρή ε, ερμηνεία. Όταν εμείς στο Πανεπιστήμιο διδάσκουμε την αρχή της επικορικότητας στους φοιτητές μας, έχουμε μια ευρύτερη αντίληψη και μια ε, πιο περιοριστική, πιο αυστηρή. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούμε πάντα την αυστηρή, την περιοριστική. Άρα η αναλογικότητα ή ακόμα και η βάση της εκχώρησης των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων δεν συζητούνται ούτε αμφισβητούνται από τα εθνικά κοινοβούλια. Νομίζω θα πρέπει να διευρύνουμε το πρίσμα μας ε, και να επιτρέψουμε και τα εθνικά κοινοβούλια όταν κάνουν τις αιτιολογημένες εκθέσεις τους όταν γνωμοδοτούν ε, με αυτόν τον τρόπο να το εξετάζουν. Νομίζω ότι αυτό θα συγκρουστεί με την άποψη νομική νομικής ακόμα και του Κοινοβουλίου, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω ακούσει κάποιους εμπειρογνώμονες εδώ, ε, ε, εγνωσμένου κύρους και διάσημους, να λένε ε, γιατί η αρχή της επικορικότητας και εκχώρηση είναι νομικά θέματα, ενώ η επικορικότητα είναι πολιτικό ζήτημα και τα εθνικά κοινοβούλια δεν δικαιούνται να εξέλθουν του στενού πλαισίου της επικορικότητας νομίζω θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Και λέγοντας όλα αυτά, θυμίζω ότι σε όλες τις ομοσπονδίες παντού όπου υπάρχει ολοκλήρωση υπάρχει και μια συνταγματική εξέλιξη. Και χωρίς αυτή την ερμηνεία, την εξελικτική, τη συνταγματική, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Στις ΗΠΑ Πολιτείες θα είχαμε apartheid και δουλεία ακόμα, αν δεν υπήρχε ευρεία ευέλικτη ερμηνεία και πώς να το πω κινούμενη εν πάση περιπτώσει ε, ε, των νόμων και των διατάξεων. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο εξετάζω στην έκθεσή μου. There Δεύτερον, υπάρχει ε, μια μαζική κίνηση, κινητοποίηση υπέρ της πράσινης κάρτας λέει ότι δεν υπάρχει βάση στη συνθήκη συνταγματική. Δεν το πιστεύω αυτό. Θα μπορούσε να είναι κάτι άτυπο. Βέβαια με κάποια πειθαρχία και με κάποια συγκράτηση και προσοχή. Έχουμε εντοπίσει έναν αριθμό η ταυτοποίηση κρατών και κοινοβούλιων που θέλουν να κάνουν αυτή την πρόταση. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι μια αντίστροφη κόκκινη κάρτα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι ε, καταργείται νομοθεσία ή κυρώνεται που υπάρχει, αλλά για πρόταση για νέα νομοθεσία. Mm-hmm. Εδώ νομίζω είναι ευρεία η συνένεση να ανοίξει νομιζω ειναι ευρια η πόρτα, η συζήτηση ή το παράθυρο, τι θέλετε, αλλά γνωρίζουμε βεβαίως ότι με πάρα πολύ άτυπο τρόπο αυτό ήδη είναι δυνατό. Διότι δεν υπάρχει κανένα εθνικό κοινοβούλιο που να απαγορεύεται να κάνει προτάσεις και από εκεί και πέρα μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει ή όχι. Αυτό όμως που θα θέλανε μάλλον είναι ότι όταν κάνουν μια πρόταση που συνυπογράφουν ξέρω εγώ 4, 5, 6 εθνικά κοινοβούλια τουλάχιστον να έχουν το δικαίωμα να τους δοθεί μια απάντηση τεκμηριωμένη. Για ποιο λόγο δεν ακολουθήθηκε η πρότασή τους. Αυτό ζητάνε. Έτσι, αυτή θα ήταν μια άτυπη πράσινη κάρτα. Το θέμα τώρα της κόκκινης κάρτας. Δεν θα μπω, δεν μπήκα πάρα πολύ σε λεπτομέρειες, διότι στην προσωπική έρευνα που έκανα σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια δεν υπάρχει πουθενά ενδιαφέρον για κόκκινη κάρτα. Λένε εδώ δεν δουλεύει η πορτοκαλί. Η κόκκινη κάρτα είχε να κάνει κάπως με το δημοψήφισμα για το Brexit και εξαφανίστηκε τελικά από τις αξιώσεις ή τις διεκδικήσεις των εθνικών κοινοβούλιων. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταγράψουμε αυτή τη συνέντευξη και να πούμε ότι δεν τίθεται πια αυτό το θέμα. Δεν είναι διεκδίκηση των ε, κοινοβουλίων, των εθνικών ή έτοιμα. Θέλω να επεκταθώ λίγο παραπάνω σε ένα θέμα, αλλά θα εξαρτηθεί αυτό από το μέγεθος της έκθεσης και των αριθμών των χαρακτήρων που έχουμε είναι να αναπτυχθεί το σύστημα IPEX που είναι τρόπος ενημέρωσης των Εθνικών Κοινοβουλίων και δικός μας. Είναι πολύ καλές ιδέες ε, που ε, έχει προτείνει το Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο το IPEX και να προχωρήσουμε. Είναι τεχνικό εργαλείο και καλό θα ήταν να το υποστηρίξουμε διότι θα μπορούσε να βελτιώσει τη πολιτική δυνατότητα διαλόγου που έχουμε. I also like to say that εδώ θέλω να τονίσω ότι ο πρόεδρος Μακρόν Πρώτη να γίνουν κάποιες δημοκρατικές συνελεύσεις άτυπες για το μέλλον της Ευρώπης. Το υιοθέτησε και ο πρόεδρος Γιούνκερ. Ίσως καλό θα ήταν να το αναφέρουμε και εμείς στην έκθεσή μας. Κάτι άλλο που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι να περιλαμβάνονται και απόψει μιοψηφία ή αποκλίουν τι απόψει στην μειοψηφία ή αποκλίνουσες αποψει στην αιτιολογημένη γνώμη των κοινοβουλίων. Σήμερα η μονολυθική. Ε, στέλνει κάθε βουλή την άποψή τη. Αλλά για να έχουν ίση εκπροσώπηση ε, με τις κυβερνήσεις θα πρέπει να αναφέρεται και η μειοψηφία. ας πούμε η άποψη της μειοψηφίας στη Σλοβακία μπορεί να είναι άποψη πλειοψηφία στην Ιρλανδία και έτσι να δημιουργηθεί και ε, μια ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ευρωπαϊκό εκλογικό σώμα, δήμος. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα τα κοινοβούλια να εγγράφουν στις εκθέσεις τους και στις νομοδοτήσεις και τις αποκλίνουν απόψη στη θέση της μειοψηφίας. Νομίζω θα ήταν χρήσιμο. Τέλος, έχουμε τη διοργανική συνεργασία όπου περιγράφονται όλα τα μέσα και τα εργαλεία που διαθέτουμε, ΚΟΖΑΚ, διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων, διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις, επιτροπές και πάει λέγοντας. Πιστεύω ότι υπάρχουν τρεις, τέσσερις, πέντε πολύ καλές προτάσεις στην έκθεση που μόλις παρουσιάστηκε από την υπηρεσία ερευνών και καλό θα ήταν να τις συμπεριλάβουμε στην επίσημη έκθεση. Αλλά και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να πλουστεύσουμε τις δομές του διακοινοβουλευτικού διαλόγου. Δηλαδή να προσπαθήσουμε πραγματικά να έχουμε ένα μοντέλο συνεργασίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με Εθνικά Κοινοβούλια για να υπάρξει κάποια ομοιογένεια στο θεσμικό μας οικοδόμημα και στο διακοινοβουλευτικό διάλογο. Και εδώ πραγματικά απευθύνω μια έκκληση. Δεν ξέρω, μπορεί να φανεί αλαζονικό από πλευρά μα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό οι κανονισμοί των Εθνικών Κοινοβουλίων να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράδειγμα, Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι τα κοινοβούλια θα είχαν πολύ μεγαλύτερο λόγο σε δημοσιονομικά θέματα αν είχαν εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των ολομελιών τους για το ευρωπαϊκό εξάμεινο για να μπορούν να κάνουν εγκαίρως τη συζήτηση νωρίς. Λένε ότι η Ευρώπη μας κλέβει τις εξουσίες μας. Δεν ισχύει αυτό. Αν αλλάξουν καμιά φορά ε, το χρονοδιάγραμμα για το πότε συζητείται ο προϋπολογισμός, μπορεί να έχουν τεράστια επιρροή στη γραμμή της κυβέρνησής τους όταν καταθέτουν τα πρώτα σχόλια ή τις πρώτες γνώμες ή τις πρώτες μελέτες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια προς το Συμβούλιο Υπουργών για το προϋπολογισμό. Και κάτι άλλο που θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα σε όλα τα κοινοβούλια ταυτόχρονα. Μια εβδομάδα αφιερωμένη σε ευρωπαϊκά θέματα, όπου ευρωβουλευτές και Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πηγαίνουν, όχι από την ίδια χώρα, ε, και να συζητούν ε, ανοιχτά και ειλικρινά ένα-δυο θέματα κάθε χρόνο, που είναι σημαντικά για το μέλλον. Αυτό πραγματικά θα ήταν μια ιδέα Ευρωπαϊκή Εβδομάδα κοινοβουλίου, με πολλές ανταλλαγές και συζητήσεις. Πώς να το πω, όλα αυτά μπορεί να είναι ευσεβείς πόθη, αλλά γιατί να σταματήσει κανείς να ονειρεύεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό, κάποιες βασικές ιδέες έτσι επιγραμματικά. Το κείμενο είναι σαφές. Είμαι απολύτως στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε για να απαντήσω σε ερωτήσεις, σχόλια κλπ. Ο Ρίτσαρτ και η Μερσέντες θέλουν να μιλήσουν. 1,5 λεπτό κατά κεφαλήν. Γιατί έχουμε καθυστερήσει και τις ψηφοφορίες. Εάν υπάρχει χρόνος. Θα γίνουν και άλλες συζητήσεις. Αν είσαστε απελπισμένος να μιλήσετε ντε και καλά, ορίστε μιλήστε. Το βασικό μου θέμα είναι ότι εστιάζουμε τόσο πολύ στην επικουρικότητα, κίτρινε, πορτοκαλί κτλ. Αλλά η επικουρικότητα είναι, δεν είναι σπάνια πρόβλημα στι νομοθετικέ προτάσει. Ε, δεν είναι συχνά πρόβλημα στι νομοθετικέ προτάσει. σπάνια είναι πρόβλημα. Γιατί καταρχά ξέρει η Κομισιόν τα νομικά τη καθήκοντα και δεύτερον, γιατί καθώ περνάει ο χρόνο, όλο και περισσότερε ευρωπαϊκέ νομοθετικέ προτάσει θέλουν να τροποποιήσουν την ισχύουσα νομοθεσία παρά να ξεκινήσουν από το μηδέν. Επομένω, είχαμε ήδη ακούσει τα επιχειρήματα ε, για το τι πρέπει να νομοθετήσουν, βασικά για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Και επιπλέον, οποιαδήποτε νομοθεσία για να υιοθετηθεί πρέπει να υποστηριχθεί από το Συμβούλιο Υπουργών με υψηλή πλειοψηφία, δηλαδή ενισχυμένη πλειοψηφία, ειδική πλειοψηφία, δηλαδή οι εθνικοί ε, υπουργοί ε, που λογοδοτούν στα εθνικά κοινοβούλια αποκλείεται να νομοθετήσουν σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο και το κάνουν μόνο αν είναι ότι πραγματικά υπάρχει λόγος Επομένω, ε, η επικουρικότητα δεν είναι πρόβλημα. Και η απόδειξη ποια είναι, ότι σε αυτά τα 7 χρόνια που ισχύει, α πούμε, σπάνια έχουμε τι κίτρινε και πορτοκαλί κάρτε. Ε, το βασικό είναι πώ τα εθνικά κοινοβούλια θα διαμορφώσουν την ουσία, όχι την επικουρικότητα. Πώ μπορούν να διαμορφώσουν τι θέσει που τελικά ε, εκφράζει το Συμβούλιο Υπουργών οι υπουργοί του. Και στην επόμενη μελέτη που θα κάνει η υπηρεσία αυτή είναι να δούμε το σκαναδικό μοντέλο, όπου δηλαδή οι υπουργοί πηγαίνουν ε, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ας πούμε, την καθήλυνα αρμόδια, πριν έρθουν στο Συμβούλιο Υπουργών, έτσι. Υπάρχει αυτή η πρακτική, έχει διαδοθεί, χρησιμοποιείται στην Ευρώπη, σε ορισμένε χώρε ναι. Ε, σε κάποιε χώρε ναι, αλλά δεν ξέρω αν διαδίδεται και στι υπόλοιπε. Μερσέντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, με το, ε, ευχαριστώ και συμφωνώ με τον Ρίτσαρτ Κόρμπετ για το θέμα της επικουρικότητας, που σπανίως αποτελεί πρόβλημα. Φυσικά, εάν προχωρήσουμε και δώσουμε αρμοδιότητες μέσω της ε, διαδικασίας που είναι εξελίξη για την ε, κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, μέσω δηλαδή της ε, διαφθομένης συνεργασίας, για την Ευρωζώνη, για τον προϋπολογισμό κτλ. Δηλαδή τότε, αν πολλαπλασιαστούν τα πεδία στα οποία παρεμβαίνουμε έτσι, με την ε, διαφθομένη συνεργασία, μπορεί να παρουσιαστούν κάποια κάζους μπέλη. Μπορεί. Πάντως, το πνεύμα της έκθεσης, θα το ξανασυζητήσουμε βεβαίως στο μέλλον, αλλά το, το πνεύμα είναι γενικά θετικό. Δεν ξεκινάει αρνητικά. Το θέμα είναι πώς θα ενσωματώσουμε τα Εθνικά Κοινοβούλια στην Ευρωπαϊκή Διαδικασία περισσότερο, ούτως ώστε να αισθάνονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και δική τους υπόθεση. Μιλάμε για μια θετική ας πούμε, συμμετοχή. Υπ' αυτή την έννοια το θέμα της πράσινης κάρτας θα μπορούσε να ενδιαφέρον. Για να γίνει μια επίσημη διαδικασία θα πρέπει να τροποποιηθούν οι συνθήκες, βεβαίως. Αλλά μπορούμε να το, βάλουμε, να το βάλουμε το θέμα αυτό στην άκρη για το μέλλον. Πάντως, στη σημερινή κατάσταση, εάν θεωρήσουμε ότι η αρχή της επικουρικότητας, όπως μας είπε ο κύριος Μαδούρο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αντίστροφα. Δηλαδή, α, κάποια κράτη μπορούν να θεωρήσουν ότι κάποιο θέμα καλό θα ήταν να έτσι περάσει περισσότερο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Όχι ότι οι ίδιοι παρετούνται εντελώ, α πούμε. Ζητούν, α πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει μια νομοθεσία, ένα νομοθετικό έργο. Υπήρξε μια τέτοια μοναδική πράσινη ε, κάρτα για να ζητήσουν μια μεγαλύτερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε, στα, στις συζητήσεις στο Παρίσι για το κλίμα. Πειραματικά λοιπόν, πιλωτικά θα μπορούσαμε να φανταστούμε διαδικασίες ε, θελοντικής πράσινης κάρτας που, χρησιμοποιούνται, χρησιμοποιούν αντίστροφα την αρχή της επικουρικότητας. Δηλαδή τα κράτη σε θέματα που θεωρούν ότι είναι αρμοδιότητά τους ζητούν παρόλα αυτά να εμπλακεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι και θετικό. Κατά τα άλλα. Να σας πω καταρχάς ότι είχα μια σκιώδη συγγήτρια που δεν μπόρεσε να παραστεί τελικά. Κρίμα είναι. Αλλά η ιδέα αυτή της εβδομάδας, η μισή εβδομάδα που είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, πολύ ενδιαφέρουσα μου φαίνεται. Γιατί κινείται και προς την κατεύθυνση που λέγαμε, δηλαδή να βοηθήσει τα Εθνικά Κοινοβούλια να συμμετάσχουν συμβουλευτικά. Αλλά εκφράζοντας την άποψή του στην ευρωπαϊκή, στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και στην νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην διαμόρφωση των πολιτικών. Ούτω ώστε όχι να υπάρχει ανταγωνισμό ανάμεσα στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά συνεργασία. ούτω ώστε να κάνουν ακόμα καλύτερα τα κράτη-μέλη αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν. Μισό λεπτό, Πάουλο, έχεις. I, I, I was only to, to, to, to say one. Απλώς κάτι θα ήθελα να πω. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Πήγα στην Αθήνα και στην Κοπενχάγη και οι Δανείοι συνάδελφοι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με το δικό του το μοντέλο. Οπότε αυτό είναι μια αλλαγή για την τελευταία φορά που πήγαμε την ΑΦΚΟ εκεί. Ήταν πάρα πολύ περήφανοι για το σύστημά του ε, και, λέγαν ότι και λένε τώρα ότι δεν δουλεύει πια και ήταν, ε, υπήρχαν, υπήρχαν μέλη του Κοινοβουλίου, ε, πρώην ευρωβουλευτέ, ε, που υποστήριζαν τη δική μας θέση και ζήτησαν μία εντολή στην Κορεπέρ. Οπότε δεν έχει... Δεν έχουν όλα τελειώσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις, τόσο περίπλοκες, που η δική μας παρέμβαση πια δεν είναι ίδια με αυτή του παρελθόντος. Άκουσα ακριβώς το ίδιο πράγμα στην Αθήνα και στην Κοπενχάγη. Ενώ είχα, είχα, πραγματικά περίμενα να ακούσω κάτι εντελώ διαφορετικό. Ήταν ε, ε, ε, πολύ διαφορετικό στο παρελθόν. Και να πω και κάτι άλλο το οποίο είπατε και είναι πολύ σημαντικό. Με την Ένωση την αμυντική ένωση έχουμε τη δυνατότητα να δούμε, ε, να να δοκιμάσουμε ένα νέο μοντέλο παρέμβασης του Κοινοβουλίου που θα είναι καινοτόμο. Θα έχουμε λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία να διερευνήσουμε αυτήν, ε, αυτό το τεράστιο δυναμικό ε, συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Μπορούμε να... Α, συγγνώμη, μισό λεπτό, μήπως έπρεπε να πω κάτι για το χρονοδιάγραμμα. Α, δεν έχουμε τη σχετική ναι. ενημέρωση. Δεν ξέρουμε καθόλου πότε θα έχουμε την έκθεσή σας. Θα σα ενημερώσω. Αύριο θα σα πω. Γιατί είχα μια, πολύ, είχα μια πολύ δύσκολη πολιτική εβδομάδα στην Πορτογαλία την περασμένη εβδομάδα και δεν πρόλαβα να το σκεφτώ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ μπορούμε τότε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον συνάδελφο από την Υπηρεσία ε, Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να δοκιμάσουμε τις κάρτες, να ελέγξουμε αν δουλεύουν ε, τα μηχανήματα. Μπορούμε λοιπόν να ελέγξουμε. You want something? Yeah, yeah, you want the Okay. Ένα e Ένας μόνο δεν έχει την κάρτα του. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε εντάξει. Ε, έχουμε 15 κάρτες που δουλεύουν, αλλά 17 ψήφισαν. Υπάρχουν κάποιες κάρτες που δεν δουλεύουν, δηλαδή. Τέλος του τεστ. Α, όχι, κάποιος μας ζήτησε να περιμένουμε. Έκθεση της ε, Mercedes Bresso, τοπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 3, υπέρ, κατά, μπορούμε να ελέγξουμε τη 3 έναρξη ψηφοφορία για την τροπολογία 3. Πέρας. Εγκρίνεται. 18. Πάμε στη συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ είναι κατά τμήματα πληροφο, ε, ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται, 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, συγγνώμη, συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 30 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία, ονομαστική, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας, εγκρίνεται 15-3. Συγχαρητήρια. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Πάμε τώρα στο Χέρολφ Άνεμας, γνωμοδότηση για το επόμενο ΠΔΠ. Δεν υπάρχουν συμβιβαστικέ, μόνο τι τροπολογίε Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 με προφορική τροπολογία, δεν διαφωνεί κανεί, υποθέτω. Οπότε ε, ψηφίζουμε τη 2 όπω τροποποιήθηκε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 4 υπέρ, συγγνώμη, 3 λέει η Πρόεδρος, 3 υπέρ, κατά, να ελέγξουμε τροπολογία 3, έναρξη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 10 προς 8. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά δεν ξέρω. Οπότε να ψηφίσουμε την τροπολογία 7 ηλεκτρονικός, έναρξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 9-9. 8 έχει αποσυρθεί. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται 11 υπέρ α όχι καταπίπτει Θέλετε να ελέγξουμε τη 10. Συγγνώμη δεν το άκουσα. Να ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικό στη 10. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 13, 3 για δύο αποχές. Η 11 καταπίπτει λόγω της 10 που εγκρίθηκε και πάμε στη 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά να ελέγξουμε τη 14 έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Οπότε εγκρίνεται η 14. Πάμε στην 20, στην επόμενη σελίδα. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 22. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 8 προς 10. 23. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος και πάλι της 23. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται 10 προς 9. Λοιπόν, καταπίπτουν πολλές και πάμε στην 27 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ. Κατά έλεγχος της 29 έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 9 προς 10. Πάμε στην 30, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 31, υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 31. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται 10 προς 9. Λοιπόν, τελική... Εγώ δεν ψήφισα στη 31. Πάμε στην τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Έναρξη. Πέρας, εγκρίνεται. 13 13 ψήφοι υπέρ, 5 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται αυτή η γνωμοδότηση. Τέλος της ψηφοφορίας για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε το απόγευμα λοιπόν στις 3 η ώρα. 3 η ώρα. Με τα Εθνικά Κοινοβούλια, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να έρθετε. Γιατί έτσι η επόμενη μελέτη του EPRS θα είναι καλύτερη αν προσέλθετε.